So, dear colleagues, ladies and gentlemen, I reopen the uh, inter-committee. Καλημέρα συνάδελφοι. Θα ήθελα να αρχίσουμε τη σημερινή συνεδρίαση ΙΝΤΑ για σήμερα. Το σημείο 14 είναι το πρώτο που θα, με το οποίο θα ασχοληθούμε. Ανταλλαγή από... Commission and I'm really glad that uh, Cecilia Malmström is here την Επίτροπο για το Εμπόριο και το Διαστρωμένο Διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα θα συζητήσουμε το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τις προϊούσες δηλαδή και μελλοντικές εργασίες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον τομέα αυτό, δεν μακρηγορώ, δίνω το λόγο στη Σεσίλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Επίσημα είναι ένας διαρθρωμένος διάλογος ο σημερινό. δηλαδή είναι η ευκαιρία που μα δίνεται να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλουμε, αλλά φυσικά επίσημα εμείς φέρουμε μια υποχρέωση να σας ενημερώσουμε σε σχέση με τα πεπραγμένα από τον τελευταίο διαρθρωμένο διάλογο και αυτό θα κάνουμε τα χαράς. Είναι αγαστή συνεργασία που έχουμε. και καλή συνεργασία από την περασμένη φορά και θα ήθελα λοιπόν να κάνω ένα απολογισμό πεπραγμένων σε σχέση με πέρσι και να σας μιλήσω για τους επόμενους μήνες. Αλλά ξανά Ξαναλέω, Πρόεδρε, μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Ήμασταν ιδιαίτερα αποσχολημένοι την περασμένη χρονιά, το ξέρετε εξάλλου και είναι πολλά τα επιτεύγματά μας. Από τον τελευταίο διαρθρωμένο διάλογο ολοκληρώσαμε δύο ε, πάρα πολύ σημαντικές συμφωνίες με τον ε, Καναδά. Πρώτα απ' όλα, ε, χτες συναντηθήκατε μαζί τους. Είναι βασικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. 99% των πρόεδρων μας ατελώς από την πρώτη μέρα θα μπαίνουν στον Καναδά και έτσι εξαγωγής ε, θα εξοικονομήσουν 470 εκατομμύρια το χρόνο και θα έχουμε επίσης πρόσβαση στις κρατικές προμήθειες σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα ε, και θα έχουμε επίσης μεγάλες ευκαιρίες για την γεωργία και τα τρόφιμα, προστασία 145 ε, κατοχυρωμένων γεωγραφικών ονομασιών γεωγραφικής προέλευσης για παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα. Ε, είναι η πιο φιλόδοξη η δεύτερη συμφωνία με το Βιετνάμ είναι η πιο φιλόδοξη που έχουμε με ασιατική χώρα και ελπίζουμε και από τις δύο πλευρές να επιτύχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη με κατάργηση των δασμολογικών φραγμών ε, θα πρέπει επίση να έχουμε ένα ισχυρό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για τα εργατικά δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ασωματωθεί στη συμφωνία και φυσικά θα παρακολουθούμε εκ του σύνα και στην εφαρμογή τη. Και οι δύο αυτές ε, συμφωνίες ε, ενέχουν και ένα άλλο πολύ σημαντικό επίτευγμα το νέο δικαστήριο, η νέα δικαιοδοτική αρχή για τη διευθέτηση των διαφορών. Είναι πολύ σημαντική η ισορροπία που επιτύχαμε. Από τη μία, τονώνουμε τι επενδύσει και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ταυτόχρονα όμω ε, ε, λειτουργούν, έχουν τη δυνατότητα οι κυβερνήσει να λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντο. Ε, αυτά εντάσσονται στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφ' εξή σε όλε τι συμφωνίε που περιλαμβάνουμε αυτή τη ρήτρα στην τίτυπα αλλά όχι μόνο και έτσι σε παγκόσμιο επίπεδο με του εταίρου μα θα διαμορφώσουμε από κοινού το νέο σύστημα σύστημα διεθνής, διεθνούς δικαιοδοτικής αρχής για την προστασία των επενδύσεων. Επίσης, χαίρομαι στο, διότι στο ΠΟΕ, στον Ναϊρόμπι, στην Διυπουργική, καταλήξαμε σε συμφωνία για την επέκταση της συμφωνίας ΙΤΑ. Μας ε, ανοίγει νέες ευκαιρίες ε, περιμένουμε την επικύρωση και ελπίζουμε να γίνει ταχύτατα, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε στο να τις νέες ευκαιρίες με την εφαρμογή της. Υπήρχαν πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα, ξεπεράσαμε και καταλήξαμε σε μια συμφωνία ε, που καταργεί την υποστήριξη προς τις γεωργικές εξαγωγές. Ε, είναι πολύ καλό αυτό για την ανάπτυξη και για την ε, προαγωγή θεμητών όρων ανταγωνισμού. Επίσης, πολύ σημαντικά βήματα έγιναν για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Την περασμένη φορά συζητήσαμε την αξιολόγηση ενός συστήματος γενικών προτιμήσεων και την κάλυψη του προγράμματος GSP-SYN. Το δημοσίευσαμε τον Ιανουάριο και το συζητήσαμε και πρώτη φορά δημοσίως και με συστηματικό τρόπο και επίσημα η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετείται για τι προσπάθειε που κάνουν οι εταίροι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη διακυβέρνηση, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπω ε, προβλέπεται και στι 27 σχετικέ διεθνεί συμβάσει ε, Στι σχέσει μα με του δικαιούχου, ε, τι χώρε εταίρου, θα πιέζουμε για πρόοδο επιτόπου. Είναι πάρα πολύ ισχυρό αυτό το έγγραφο που δημοσιεύσαμε. Επίση, έχουμε αρχές συμβόσιμες ανάπτυξη και σχετικέ ρήτρε στι νέε συμφωνίε που με τον Καναδά και το Βιετνάμ για τα ανθρώπινα ανθρώπινα δικαιώματα, για την βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος, ενίσχυση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων σε σχέση με τι εργασιακές σχέσεις, είναι ζητήματα που τονίζουμε σχέση με τους εταίρους μας. Επίσης ε, αυξάνεται η συμμετοχή της κοινωνίας των εταίρων ε, όχι μόνο για τις αποφάσεις αλλά και για την εφαρμογή αυτών. Επίσης ε, για την βιώσιμη ανάπτυξη στις διαπραγματεύσεις TTIP με τις ΗΠΑ έχουμε επίσης διαπραγματευτεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο όπου υπάρχουν υποχρεώσεις αμφοδέρων των πλευρών και τονώνεται η διατλαντική συνεργασία ούτω ώστε αυτές οι αξίες να εξαχθούν τρόπον την σε άλλες χώρες, τρίτες χώρες και νομίζω ότι θα είναι ρηξικέλευτα τα αποτελέσματα και έχουμε αναλάβει ιδιαίτερα ισχυρή δέσμευση στι διαπραγματεύσει μα, ώστε να έχουμε εφάμιλε φιλοδοξίε στον τομέα αυτά. Αυτά έχουμε πετύχει. Τι ε, έπεται τώρα. Ε, φυσικά εφαρμογή της στρατηγικής Trade for All. Ε, από πέρυσι τον Οκτώβριο αυτό μας απασχολεί, είναι προϊούσες οι εργασίες μας ε, και φυσικά έχουμε ξεκινήσει, έχουμε δρομολογήσει τις πρώτες δράσεις για την αποτελεσματικότητα, παραδείγματος χάρη διατάξεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλες τις εμπορικές μας συμφωνίες. Επίσης, ιδέες νέες εταιρικές σχέσεις για να εφαρμόσουμε καλύτερα αυτές τις συμφωνίες, ε, διότι θα πρέπει να φέρουμε βελτιώσεις ε, για την διαφάνεια, το μοντέλο TTIP. Δημοσιεύουμε το μέγιστο αριθμό εγγράφων από διάφορε διαπραγματεύσει ε, για τι ε, συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών, ΣΕΣ, και θα συνεχίσουμε τι προσπάθειε και στο μέλλον. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για τον προσδιορισμό νέα προσέγγιση για τη συμπερίληψη διατάξεων καταπολέμηση ε, τη διαφθορά στι εμπορικέ μα συμφωνίε. Αυτή την εβδομάδα είναι η εβδομάδα κεραιότητα ε, και στον ΩΣΑ, στο Παρίσι. Έγινε μια πολύ μεγάλη διάσκεψη. Ήμουν παρούσα και φυσικά, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Είναι κάτι που μπορούμε, από το οποίο μπορούμε να αποκομίσουμε πολλά ωφέλη αν κινηθούμε σωστά. Εκπλήρωση λοιπόν όλων των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει στα πλαίσια της στρατηγικής Trade for All και περιμένουμε με ανυπομονησία και τη δική σας έκθεση, ούτως ώστε να λάβουμε υπόψη και τη δική, τα, δική σας, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις. Επίσης, αν, το Δεκέμβριο αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη νέα θετική όθηση που υπάρχει από πλευρά του ΠΟΕ για να αναζωογονήσουμε τις σχέσεις μας και το ρόλο μας στον ΠΟΕ. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα σε σχέση με την Ολλανδική Προεδρία και στις 13 Μαΐου ε, ε, στο επόμενο Συμβούλιο θα το συζητήσουμε αυτό. Φυσικά τα εκκρεμή ζητήματα του γύρου της Ντόχα γιατί μόνο ο ΠΟΕ μπορεί να ασχοληθεί με ζητήματα όπως ε, εγχώρια στήριξη ή βιομηχανικές επιδοτήσεις φυσικά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Ταυτόχρονα χρειάζεται επικαιροποίηση για νέα ζητήματα. Πολλά κράτη-μέλη και πολύ και θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα μια σχετική σημαντική σύσκεψη για ζητήματα όπω ψηφιακό εμπόριο, ε, βέλτιστε ρυθμιστικέ πρακτικέ και εμπορικοί περιορισμοί. Θα θέλαμε να έχουμε πιο στοχευμένους, ε, στοχευμένες φιλοδοξίες για να ε, τις προωθήσουμε σχέσεις μας με τους εταίρους μας. Ε, σε πολυμερές επίπεδο καταρχάς και αν αυτό δεν είναι δυνατό μπορούμε να δούμε εάν μπορούμε σε ε, πολυμερές επίπεδο να ξεκινήσουμε και να ενσωματωθούν στη συνέχεια στο σύστημα ΠΟΕ αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Επίσης, διμερείς και περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες. Θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την, τον εξυγχρονισμό της ε, ΣΕΣΕ με το Μεξικό. Συναντήθηκα με τον Υπουργό αυτή την εβδομάδα και είμαστε στο τελικό χτένισμα, ώστε να ετοιμάσουμε και την εντολή που θα μας δώσουν τα κράτη-μέλη. Σε λίγες εβδομάδες θα είναι έτοιμη, ελπίζουμε. Ε, για τις διαπραγματεύσεις Mercosur επίσης ε, καθυστερήσαμε για πάρα πολύ καιρό και ο στόχος είναι να έχουμε νέες προσφορές στο πρώτο ήμιση του Μαΐου και θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή μετά το 2004. Έχουν συμβεί πάρα πολλά έκτοτε και εξακολουθούν να συμβαίνουν σε διάφορες χώρες, Mercosur Είναι καταπληκτικές ευκαιρίες που ανοίγουν έρχονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για το Μερκοσούρ. Για τις ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρική σχέσης, ε, ΣΑΝΤΙΚ και ΕΑΚ ε, προτείνεται η υπογραφή και ελπίζω να δώσει το πράσινο φως το Συμβούλιο τόσο ώστε πριν το καλοκαίρι να υπογραφούν. Ουκρανία επίσης αρχίζει η συμφωνία να ισχύει από πρώτης πρώτη ούτως ή άλλως και τώρα Συνεργαζόμαστε με την Ουκρανική κυβέρνηση ώστε να την εκμεταλλευτούμε. Φυσικά όμως συνεχίζεται η διαδικασία εφαρμογής και παρακολούθησης και το ίδιο και με την Μολδαβία και τη Γεωργία. Πρόσφατα επισκέφθηκα αυτές τις γειτονικές χώρες και αυτή την εβδομάδα κάνουμε γύρω διαπραγματεύσεων με την, την Ισία για να στραφούμε προς τους νότιους γείτονές μας και προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ ε, που έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις. Για την Ασία πριν από τα Χριστούγεννα ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις με τις Φιλιππίνες και ε, τον πρώτο γύρο, επίσημο γύρο, θα τον έχουμε ε, πολύ σύντομα εδώ στις Βρυξέλλες. Είναι η πέμπτη διμερής διαπραγμάτευση ε, με εταιρό από την Ασία. Θέλουμε, όπως και για τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ, να κινηθούμε στο ίδιο επίπεδο. Είναι ραγδαία αναπτυσσόμενη η οικονομία της χώρας και θέλουμε να μην χάσουμε την ευκαιρία του, της αγοράς του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων καταναλωτών. Ε, και τέλος, ε, με ο Πρόεδρος ε, και ο Υπουργός Εμπορίου της Ινδονησίας θα συναντηθούν με ένα μεγάλο κλιμάκι από την Ινδονησία με τον Πρόεδρο Γιούνκερ σήμερα. Ελπίζουμε να αποφασιστεί η δρομολόγηση των διαπραγματεύσεων και με την Ινδονησία. Έχουμε ε, τι περασμένε εβδομάδε ε, κάνει πάρα πολύ εντατικέ προετοιμασίε, Είναι πολύ ιδιαίτερα προστατευτικό το σύστημα τη χώρα και τώρα ανοίγονται και θέλουν ε, να αναλάβουν μια δέσμευση στις διμερείς σχέσεις με την ΕΕ. Είναι πολύ φορτωμένο το θεματολόγιο μα Έχουμε το, την Ιαπωνία, την επενδυτική συμφωνία με την Κίνα. Όλα αυτά τρέχουν ταυτόχρονα. Επίσης, νομοθετικές προτάσεις. Ε, την επεξεργα... επεξεργαζόμαστε σε συνεργασία με και το Συμβούλιο. Ελπίζω πραγματικά να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των συνομοθετών ε, για τα ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες. Ε, ξέρω ότι ε, αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα και εμείς το ίδιο είχαμε δύο τριμερείς διαλόγους. Περιμένουμε τώρα το Συμβούλιο και το Πρόεδρο Λάγκια και πολλούς από εσά να βρείτε μία κοινή γραμμή και στο Συμβούλιο ελπίζουμε να προχωρήσει το θέμα ώστε πριν το καλοκαίρι να έχουμε και σε αυτό το τομέα εξελίξεις. Επίσης, το εργαλείο για τις κρατικέ προμήθειες σε διεθνές επίπεδο επίπεδο εγκρίθηκε εδώ αναθεωρημένη πρόταση και σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ελπίζουμε και εκεί να σημειωθεί η πρόοδος. Εξυγχρονισμός των εργαλείων ε, προστασίας του εμπορίου, από ό,τι έμαθα, το συζήτησατε πρόσφατα εδώ, έχει μπλοκαστεί διαδικασία στο Συμβούλιο, πάντως ε, χρειάζεται αυτή η συζήτηση, πρέπει να γίνει και ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα είναι σε θέση να το συζητήσει στην ε, στο επόμενο Συμβούλιο, γιατί έχουμε και το πρόβλημα στο Χάλιβα. Ε, το Μάιο, γιατί ξέρω ότι θα με ρωτήσετε πολλά γι' αυτό, ε, Κίνα και έρευνε ε, για τα μέτρα αντι-dumping. δεν έχει το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ε, αυτό που εξετάζουμε είναι πώς ακριβώς ε, θα υπολογίσουμε τα μετρα αντι anti-dumping και τις ε, σχετικές έρευνες που γινόνται για κάποιες ερήτρες του πρωτοκόλ προσχώρησης του ΠΟΕ που εκπνέει το Δεκέμβρη για την Κίνα. Εξετάζουμε λοιπόν πολύ προσεκτικά αυτό το ζήτημα, το ξέρετε. Χτες ε, το βράδυ ε, έληξε και η προθεσμία για τη δημόσια διαβούλευση. 5.000 απαντήσεις μου είπαν οι συνεργάτε μου ότι λάβαμε και αυξανόταν γεωμετρικά ο ρυθμός τους τελευταίες δύο ημέρες. Πρέπει να τι αναλύσουμε φυσικά. Έγιναν και εκδηλώσεις με του εμπλεκόμενου φορεί stakeholders, ε, για να ακούσουμε ε, τις απόψεις τους για αυτό το ζήτημα και φυσικά θα καταρτήσουμε ένα συνοπτικό πίνακα και θα δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα Τη ε, δημόσια διαβούλευση. Επίση, λεπτομέρειε των επιπτώσεων μιασδήποτε αλλαγή που ενδεχομένω ε, γίνει, το ίδιο και για την ανάπτυξη και τι θέσει εργασία για την οικονομία και ε, ενδεχομένω χρειάζονται μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων των νέων εργαλείων προστασία των εμπορικών συναλλαγών. Συνεχίζεται η διαδικασία και ελπίζω να έχουμε ολοκληρώσει τον Ιούνιο, ώστε να αρχίσουμε την συζήτηση με, του υπόλοιπου επιτρόπου. Ε, πολύ ασχολούνται με αυτό το ζήτημα ε, και κάνουμε ε, ανοιχτές συζητήσεις και προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη ε, όλες τις απόψεις. Για την ευημερία μας χρειαζόμαστε ανοιχτές αγορές, αλλά όχι μόνο, χρειαζόμαστε και αποτελεσματικά εργαλεία προστασίας του εμπορίου και επ' αυτή της βάσης θα λάβουμε την απόφασή μας συνυπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους. Να, κάποια λίγα ζητήματα που επεξεργάζουμε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα ξέχασα κάποια, θα μου τα θυμίσετε εσείς ευχαριστώ πάντως για την σημερινή ευκαιρία και προσβλέπω στην σημερινή μας συζήτηση. Ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσω τη συζήτηση, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεν είναι μια συνήθις διαδικασία ερωταπαντήσεων, είναι μια συνεδρίαση στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου, όπως είπε και η Επίτροπος. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με τις προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας και να συζητήσουμε και το επερχόμενο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να συνοψίσουμε όσα θα υποθούν, να το συζητήσουμε με τις πολιτικές ομάδες και να το αποστείλουμε στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, η οποία θα υποβάλει το αποτέλεσμα των ε, διαλόγων αυτών από όλες τις επιτροπές στη διάσκεψη των Προέδρων, ούτως ώστε να υπάρξει θέση, ελπίζω, του Κοινοβουλίου μετά το καλοκαίρι για το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να δώσω πρώτα το λόγο λοιπόν στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και κατόπιν στους άλλους συναδέλφους. Σας παρακαλώ να μην υπερβείτε τα τρία λεπτά για να υπάρξει επαρκής χρόνος και για συζήτηση και να μπορέσουν να πάρουν το λόγο όσοι θέλουν να συμμετάσχουν. Κασπάρι πρώτος, ΕΛΚ. Αγαπητή κυρία Επίτροπε, αγαπητή Σεσίλια, νομίζω ότι παρουσιάσατε πολύ καλά το ότι έχουμε πολλές επιτυχίες στα θέματα εξωτερικού εμπορίου, χάρη και στη δική σας προσπάθεια για τον ΠΟΕΣ, τον Ναϊρόμπι, για παράδειγμα. Αν δεν ήξερα ότι ε, χρειάζεται διερμηνία από τα γερμανικά στα γερμανικά. Λοιπόν, τι έλεγα. Λοιπόν, υπάρχουν επιτυχίες. Είναι μεγάλο βήμα αυτό που συνέβη για τον ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι. Είναι τεράστιο βήμα η συμφωνία ΣΥΤΑ και η συμφωνία με το Βιετνάμ. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Είναι επίσης, ε, επίσης μεγάλη η δική σας ε, επιτυχία ότι προχωράνε οι διαπραγματεύσεις Μέρκοσουρ και αλλού. Αλλά ανησυχώ για ορισμένα θέματα που δεν είναι εκτός ε, αλλά εντός της Ευρώπης είπατε ότι υπάρχουν πολλά νομοθετικά θέματα που δεν προχωρούν για παράδειγμα η μεταρρύθμιση του TDR υπάρχουν και άλλα νομοθετικά θέματα βλέπω ότι υπάρχει μια νέα πρόταση της Κομισιόν ε, η οποία ε, δεν προχωράει στο Συμβούλιο ενώ προχωράει, ενώ προχωράει βέβαια στο Κοινοβούλιο για τα ε, ορυκτά σε περιοχές συγκρούσεων επίσης γίνονται συζητήσεις αλλά δεν γίνεται τίποτα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε λοιπόν ούτως ώστε το θέμα του ότι το Συμβούλιο έχει μπλοκάρει όλα τα νομοθετικά θέματα να το υπερβούμε για τη Σιγκαπούρη. Κάποια στιγμή θα επανέλθει το θέμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για αυτή τη συμφωνία. Έχουμε καταλήξει στις διαπραγματεύσεις, αλλά για την προστασία των επενδύσεων για, την Βιετνάμ, για το Βιετνάμ και τον Καναδά έχουμε αποφασίσει διαφορετικά. Έχει υπόψη της τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν, ούτως ώστε να μην χάσουμε χρόνο, τι μπορούμε να φτιάξουμε στη συμφωνία με την Σιγκαπούρη, θα αρχίσουμε τη διαδικασία επικύρωσης ή θα κάνουμε συμπροματικές διαπραγματεύσεις. Και το τρίτο σημαντικό θέμα, η οικονομία της αγοράς. Εφόσον είναι διαθρωμένος ε, διάλογος, είναι σίγουρα μία από τις κύριες προτεραιότητες για το δεύτερο εξάμεινο. Είναι σημαντικό για την ομάδα μας και μετά τον ερχόμενο Δεκέμβριο να έχουμε ένα ε, αποτελεσματικό μέσο anti-dumping. Να έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντά μας ενώπιον του ΠΟΕ. Είναι δύσκολο λοιπόν, επειδή γίνεται συζήτηση για αυτό το θέμα, να παραμείνουμε αδρανείς. Είπατε λοιπόν ότι θα αποτιμήσετε τα αποτελέσματα του δημοσίου διαλόγου τον Ιούνιο. Αλλά πώς είναι το χρονοδιάγραμμά σας συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μπορούμε να πούμε στους πολίτες μας που ανησυχούν τι θα γίνει μετά τον Ιούνιο για την χορήγηση ή όχι καθεστώτος οικονομίας της αγοράς για την Κίνα και να έχουμε δυνατότητα να χρειαστεί να προωθήσουμε και έγκαιρα την νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστώ. David Martin για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Και άλλοι συνάδελφοι έχουν ερωτήσει, Θα επιχειρήσω να είμαι σύντομος για την ε, πολυμερή προσέγγιση Χαίρομαι ότι συνεχίζετε, να τονίζετε τη δέσμευσή σας για την πολυμερή προσέγγιση και δεν συμφωνείτε με αυτούς που λένε ότι η ΝΤΟΑ έχει πεθάνει. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε για μια πολυμερή προσέγγιση. Σας στηρίζουμε λοιπόν πλήρως και ήθελα να το πω. Και θα πρέπει στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου για το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν να αναφερθεί αυτό. Δεύτερον, με βάση και αυτά που μόλις είπε ο Ντάνιελ, αλλά και εσείς για τα αμυντικά μέσα στην, για τα μέσα εμπορικής άμυνας. Είπατε ότι δεν θα είναι στην ημερήσια διάταξη το Μάιο του Συμβουλίου. Εμείς θα πιέσουμε ως Συμβούλιο. Και ξέρω ότι κατηδίαν κάνετε και εσείς ό,τι μπορείτε. Αλλά νομίζω ότι χωρίς να θέλω να δημιουργήσω προβλήματα στις σχέσεις μας με το Συμβούλιο ή την Προεδρία ή με κάποια κράτη-μέλη. Ε, πρέπει κάτι να κάνει η Κομισιόν γιατί πολλά κράτη-μέλη ε, δρούν υποκριτικά. Κρίνουν και επικρίνουν την Κομισιόν ότι αργεί να υποβάλει προτάσεις για αυτά τα μέσα εμπορική άμυνα, αλλά μετά κολυσιεργούν. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να κάνουμε. Υπάρχει κολλησιεργουν πρεπει οπωσδηποτε κατι να πρέπει να μπει στην ημερήσια διάταξη του Μαΐου. Θα ήταν πραγματικά σοβαρή παράληψη αν δεν γινόταν αυτό. Κάτι άλλο που δεν έχουμε συζητήσει, αν δεν κάνω λάθος, είναι η δυτή χρήση. Και νομίζω ότι το έχουμε ξεχάσει αυτό κάπως, γιατί είναι σχεδόν δύο χρόνια από τότε που τα θεσμικά όργανα έχουν ασχοληθεί και έχουν κάνει μια δήλωση για το θέμα αυτό. Οποτεδήποτε έχουμε άλλα προβλήματα σημαντικά όπως ε, η τρομοκρατία, η εγκληματική δραστηριότητα που εξαπλώνονται. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό πρέπει να ενημερώσουμε τους κανόνες μας για την διτή χρήση. Διερωτώ με πότε η Κομισιόν θα κάνει πρόταση από αυτού. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τα σχόλια που κάνατε. Ήδη καλύπτουν κάποια θέματα που ήθελα και εγώ να θέσω. Το πρώτο ήταν φυσικά η Ασία και πόσο σημαντικό είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας, ιδιαίτερα με τις αναδυόμενες αγορές. Ε, χάρηκα που αναφερθήκατε στην Ινδονησία και όπως και ο συνάδελφος ε, κύριος Κασπάρη έχει σημασία στην περιοχή αυτή και η Σιγκαπούρη. Πρέπει λοιπόν να σημειωθεί πρόοδος. Ε, έχετε χρονοδιάγραμμα λοιπόν γι' αυτό και κάνετε κάτι για να, το, για να επιταχύνετε την εξέταση του θέματος αυτού. Θέλω να μην το ξεχάσουμε, να το προωθήσουμε το θέμα αυτό. Επίσης, θέλω να ρωτήσω για την Ταϊβάν μπορούμε να προωθήσουμε την συμφωνία επενδύσεων του Ταϊουάν συνδέεται με το θέμα της Κίνας ε, γιατί με την Κίνα βέβαια έχουμε το θέμα των συζητήσεων για το καθεστώς οικονομίας της αγοράς μήπως θα μπορούσε να ε, λήξει η συμφωνία μας με την Ταϊουάν προηγουμένως και τι γίνεται με την Ινδία μετά τη συνάντηση κορυφής που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες υπήρξε κάποια κίνηση από την πλευρά τους να δημιουργήσουμε έναν ε, τακτικό διάλογο για να συζητήσουμε θέμα όπως ε, τα αυτοκίνητα, ε, είναι κοινοβρεματόδη, υπάρχει κάποια κίνηση σε επίπεδο υπουργών. Χαίρομαι για την συμφωνία με το Μεξικό. Επίσης, ε, να εστιάσω περισσότερο στο ότι καθυστερούμε να καταλήξουμε σε συμφωνίες αλλά μετά αργεί πολύ και ο νομικός έλεγχος, η νομική επαλήθευση, legal scrubbing, ιδιαίτερα επειδή κάποια συμφωνία κατέληξε και υπεγράφει εντός έξι μηνών. Για την Νότια Κορέα ένα χρόνο, ε, ένα χρόνο και 7 ε, μήνες για το ΣΥΤΑ, 18 μήνες για τη Σιγκαπούρη. Νομίζω ότι επειδή υπάρχει τόση διάθεση για εμπόριο, πρέπει και εμεί ε, να επιταχύνουμε τι διαδικασίε μα, να μειώνεται ο χρόνο μεταξύ κατάληξη διαπραγματεύσεων και υπογραφή των συμφωνιών. Αλλά θέλω να χαιρετήσω την εργασία που γίνει για το TTIP, για τι μικρομεσαίε και νομίζω ότι άκουσα σωστά ότι θέλετε να υπάρχει κεφάλαιο για τι μικρομεσαίε στι μελλοντικέ εμπορικέ συμφωνίε. Οπωσδήποτε η ομάδα μου θέλει αυτό να συμπεριλαμβάνεται σε τέτοιε συμφωνίε. Ευχαριστώ, η Μαρίτια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Να συνεχίσω από όλα τα σημαντικά σχόλια που έκανε η συνάδελφη. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπάρχει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα και επί τον οποίο αναζητούμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι φιλοδοξία μιας ε, πιο ολοκληρωμένη ατζέντα για το εμπόριο, που έχει συγκεκριμένε αξίε και θέλει να έχει εμπόριο για όλου, μπορεί να υλοποιηθεί με τι δυνατότητε που έχετε τώρα στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Συζητήσαμε χθε ε, το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τι πιθανέ προσθήκε ή προσαρμογέ που θέλουμε να κάνουμε και ήθελα να θέσω το γεγονό ότι υπάρχουν πολλέ προσδοκίε, όχι μόνο σε θέματα διαφάνεια, αλλά όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών, ε, οι πορευόμενοι θέλουν να εισακουστούν. Και δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα προσδοκία επικοινωνίας και προσέγγισης και ε, συζήτησης με τους ε, ανθρώπους αυτούς. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν οι δυνατότητες στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, αν χρειαστεί. Δεύτερον, συμφωνώ απολύτω με αυτό που είπε ο Ντάνιελ Κασπάρη για τη αδιέξοδο στο Συμβούλιο σε πολλά ζητήματα. Είναι ανησυχητικό αυτό. Και λόγω αυτού θα ήθελα να ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε κάποια περισσότερα για τις φήμες που ακούμε για το ενδεχόμενο πρόεδρος Ομπάμα να ε, προτείνει ε, μία περιορισμένη TTIP ε, στη σύνοδο που θα κάνει στις επόμενες ημέρες με κάποιους από τους ηγέτες εδώ στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι αυτό δεν θα ήταν καλό γιατί τα θέματα για την πρόσβαση στις αγορές και τις δημόσιες συμβάσεις δεν έχουν ελοποιηθεί και ήταν θέματα τα οποία ανησυχούν την Ευρώπη ήδη. Δεν νομίζω ότι θα προκύψει λοιπόν κάτι καλό από πολιτική σκοπιά σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης, θα ήθελα να σταθώ στην ανάγκη για επικαιροποίηση του κανονισμού για τα προϊόντα διπλής χρήσης. Υπάρχουν ε, προβλήματα πρακτικά. Ε, υπάρχουν προϊόντα τα οποία αναπτύσσονται λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας πολύ γρήγορα και είναι μικρότερα, φθηνότερα, ε, πιο εύχριστα και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ε, ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας. Είδαμε ότι η Ιταλία ανακάλεσε την άδεια για πωλήσει εκτός Ευρώπης για μια Ιταλική επιχείρηση που κατηγορήθηκε ότι πουλά λογισμικό σε απολυτερχικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο, κάτι το οποίο δεν είναι καν ε, νόμιμο μάλλον. Εάν λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε τέτοια πωλήσει και δεν υπάρχει λογοδοσία και διαφάνεια, υπάρχει πρόβλημα με τον κανονισμό. Επισημαίνω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει κάποια πρόοδο στο σημείο αυτό. Ε, θα σταθώ σε αυτό γιατί πρέπει να δώσουμε και στους άλλους αδέλφους τη δυνατότητα να παρέμβουν. Ο Χέλμουντ Σόλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Μάλστρομ. Κάποια σχόλια για ορισμένα που ήδη υπόθηκαν και κάποια για τα κεντρικά θέματα που έχετε θέσει και κάποια για το μέλλον. Για την εμπορική σας στρατηγική ε, ασχοληθήκατε ιδιαίτερα στο δίκαιο εμπόριο. Συμφωνώ, πρέπει να επιμείνουμε. Πώς θέλουμε να υπάρξει δίκαιο εμπόριο και εντός των χωρών μας και σε επίπεδο ένωσης και εκτός Μόνο έτσι θα γίνει κάτι ουσιαστικό και πραγματικό απτό για τους ε, πολίτες μας. Είπατε βεβαίως, πρώτα απ' όλα πω, ε, ναι, θέλουμε πολυμερή προσέγγιση, αλλά το θέμα είναι τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Όταν κάνουμε την απαρίθμηση, διαπιστώνουμε ότι οι διμερείς συμφωνίες και προσεγγίσεις είναι πολύ περισσότερες από τις πολυμερείς. Άρα και για το επόμενο πρόγραμμα σας πώς θα περιλάβει ενισχυμένη αναφορά στην πολυμερή προσέγγιση στα διάφορα κεφάλαια, στα διάφορα θέματα που θέλετε να διαπραγματευτείτε. Δεύτερον, χθες αναφερθήκαμε στον προϋπολογισμό και τις πολιετής προοπτικές. Πρέπει να πω ότι πρέπει να ενημερώσουμε τα στοιχεία μας για να δούμε πού έχουμε λιγότερα, λιγότερα έσοδα λόγω του ότι μειώνονται για παράδειγμα οι δασμοί άρα θα έχουμε λιγότερα έσοδα και με τι έσοδα θα τα αντικαταστήσουμε για να ενισχυθεί η Ένωση. Εάν λόγω της πολιτικής μας δεν υπάρχουν πλέον καθόλου ε, ε, δασμοί δεν θα έχουμε επαρκή έσοδα, επαρκείς ίδιους πορου Τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν, εσει ε, και οι άλλοι επίτροποι οι οποίοι είναι αρμόδιοι για αυτά τα θέματα, πώ θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό. Έχετε μια στρατηγική για το πώ ε, θα αντιμετωπίσετε τις επιπτώσεις ε, τη πολιτική εμπορίου, τη εμπορική πολιτική σε άλλα θέματα. Πρέπει να θέσουμε το θέμα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, για παράδειγμα, ή κάποια άλλα. Έχουμε τα στοιχεία από το Panama Leaks. Έχουμε τα στοιχεία για το φορολογικό dumping. Υπάρχουν πολλοί τομεί του οποίου απλώ θέλω να θίξω ακροφυγός, ότι πρέπει να τους λάβουμε υπόψη ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μια σαφή νομοθετική βάση για να αποκαταστήσουμε την κατάσταση των εσόδων μας. Ναι, άλλο θέμα τώρα. Βεβαίως ε, η οικονομία της αγοράς για την Κίνα τεράστιο θέμα. Το Μάρτιο στην Ολομέλεια θέλαμε με μια διμερή συμφωνία να αποκαταστήσουμε την ε, ανταγωνιστικότητα των σχέσεων μας με την Κίνα, να αντιμετωπίσουμε το θέμα του ντάμπινγκ κτλ. Να μην υπάρξει λοιπόν σύγκρουση. Υπάρχουν πολλά θέματα. Τι θα γίνει με τη Ρωσία, τι θα γίνει με τη διαφθορά στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με τις οποίες έχουμε εμπορικές συμφωνίες, Ουκρανία και Μολδαβία. Η Μολδαβία, σύμφωνα με την εκτίμηση του πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποτύχει το κράτος, έχει καταρρεύσει. Ευχαριστώ, λέει ο Αυτοί ήταν οι συντονιστές. Τώρα έχουν ζητήσει άλλοι 11 συνάδελφοι το λόγο και θα είμαι λοιπόν πολύ αυστηρός όσον αφορά την τήρηση του χρονικού όριου. Κύριο κύριος Μπούχνερ, πρώτος. Α, ωραία, ωραία. Ε, α, και εσείς θέλετε. Οπότε είναι 12. Δεν επιτρέπεται άλλος. 12. Πρώτη είναι η Darling. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Να σας πω καταρχάς ότι χαίρομαι για τη δέσμευση που αναλάβατε ως Επίτροπος το 2014 για κοινοβουλευτικό έλεγχο και ε, συμμετοχή στο Κοινοβούλιο και συνομιλίες με το Κοινοβούλιο. Έχουμε δει μεγάλη πρόοδο, κυρίως όσον αφορά το κοινοβουλευτικό έλεγχο, τη διαφάνεια και την αυξημένη δημοκρατία στην ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική. Θεωρώ ότι είναι θετική αυτή η πρόοδος και πρέπει να την προωθήσουμε. Φαντάζομαι ότι θα γνωρίζετε ότι στα πλαίσια του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν ε, ε, θέματα περί δημοκρατικού ελέγχου και πώς ε, εξελίσσεται η εμπορική πολιτική και υπάρχουν όλοι αυτοί οι μύθοι και ψεύδοι ορισμένες φορές που διαδίδει η εκστρατεία υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν μια δήλωση από πλευρά σας για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπόλογη στους πολίτες της όσον αφορά την εμπορική της πολιτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση δρά προς το συμφέρον των πολιτών της ε, στις διαπραγματεύσεις της. Η επέκταση της διαφάνειας που είδαμε στι ε, ε, συμφωνίες ε, και στις διαπραγματεύσεις για την TTIP και την TISA δείχνουν ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν αυτό είναι στα μελλοντικά σας σχέδια. Τώρα, Όσον αφορά τη δημοκρατική συμμετοχή και το δημοκρατικό έλεγχο, ε, ένα θέμα το οποίο απασχολεί είναι η προσωρινή εφαρμογή των συμφωνιών. Και έχουμε δει αρκετά σχόλια για το πώ θα αντιμετωπίζονται μελλοντικέ εμπορικέ συμφωνίε όσον αφορά την προσωρινή του εφαρμογή. Από νομική σκοπιά ξέρουμε ότι οι υπουργοί μα μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν προσωρινά μία συμφωνία πριν ε, ε, ψηφίσει επί τη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό περιλαμβάνεται στη συνθήκη. Το έχει προσυπογράψει και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά ε, ε, θα θέλαμε κανονικά να ψηφίζει το Κοινοβούλιο πριν υπάρξει οποιαδήποτε προσωρινή εφαρμογή. Ε, δεν ξέρω κατά πόσον θα συνεχίσει αυτή η πρακτική. Ε, εσείς είπατε ότι δεν θέλετε να συνεχιστεί, αλλά ακούμε κάποιες αμφιβολίες από κάποιους ε, ε οι οποίοι κάνουν εκστρατείο και από κάποιες ε, πλευρές ότι θα μπορούσε να υπάρξει προσωρινή εφαρμογή της ΣΥΤΑ ή της ΤΙΤΙΠ πριν ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πραγματικά λοιπόν θα ήθελα δέσμευση από εσά σήμερα, στεναρή δέσμευση, ότι δεν ε, θα εφαρμοστεί καμία συμφωνία προσωρινά πριν ψηφίσει από αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρωθεί εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, κυρία Μίνερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω από αυτά που είπε η κυρία Κερτον Ντάρλινγκ. Διότι έθεσε το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων. Ξέρουμε ότι υπάρχει δήλωση ενός Ινστιτούτου που λέει ότι το δικαίωμα για νομοθεσία δεν μπορεί να μείνει ε, Στη χώρα μου υπάρχει μία συζήτηση. Η Επιτροπή ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είπε σήμερα ότι οι αγρότες ε, θα αντιταχθούν στη TTIP. Υπάρχουν μεγάλες αντιρρήσεις για αυτές τις εμπορικές συμφωνίες και κινητοποιείται η κοινωνία. Εχθές η Καναδή Υπουργός, η κυρία Φρίλαντ που ήταν εδώ, μας είπε ότι η συμφωνία θα ξεκινήσει να ισχύει από αρχές του έτους, δηλαδή πριν προλάβουν τα κράτη-μέλη να τη συζητήσουν. Έχουμε δει ότι στην περίπτωση της Ουκρανίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει ότι η συμφωνία μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται προσωρινά επαόριστον νόμος. Και εγώ θέλω πρώτα να υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία στα κράτη-μέλη και πριν κυρωθεί ή αποφασίσει ένα κοινοβούλιο επί της συμφωνίας να μην τίθεται σε ηχή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας κύριε Επίτροπε και σας ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία πολύ συγκεκριμένα θέματα. Το ένα αφορά τη σχέση με τη Λατινική Αμερική από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει ανταλλαγή προσφορών με τη Μερκοσούρ ε, στα μέσα Μαΐου και θεωρώ ότι είναι καλή είδηση αυτή, αλλά λόγω της πολιτικής αστάθειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βραζιλία θα ήθελα να ξέρω ε, τι κινδύνου βλέπετε εσείς ε, αν μπορεί να συνεχιστεί ομαλά η διαδικασία και τι ε, ε, βλέπετε ε, αν μπορούμε να αποφύγουμε αυτά που είχαν συμβεί στο παρελθόν και να έχουμε μια επιτυχή διαδικασία. Για την περίπτωση του σημερινού. Όλοι συνειδητοποιούμε ότι εάν δεν τεθεί σε εφαρμογή συμφωνία με το Εκουαδόρ, την προσχώρηση στη συμφωνία με την Κολομβία και το Περού δηλαδή και για τον Ισημερινό, θα περιπλακούν πολύ τα πράγματα διότι σταματάει να ισχύει το GSP+. Plus Και επομένως θα περιπλακεί, ε, είναι συγγνώμη, πιο περίπλοκη η κατάσταση στον Ισημερινό και λόγω του σεισμού. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι θα μπορέσει να γίνει ώστε να μπορέσουμε να καθησυχάσουμε τους ε, κατοίκους του σημερινού για να μπορέσουμε να σταθούμε και στο ύψος των περιστάσεων και να κυρώσουμε τη συμφωνία για να τεθεί σε ισχύ για να μπορέσουμε να βιώσουμε και την οικονομία τους. Και για να ολοκληρώσω και με τη Λατινική Αμερική, τι χρονοδιάγραμμα έρχεται για τον εξυγχρονισμό της συμφωνίας με τη Χιλή. Δεύτερον, για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των ε, συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί. Νομίζω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να αυξηθεί ο αριθμός των συμφωνιών που υπογράφονται με τρίτες χώρες, αλλά αν δεν συνοδεύεται και από αυτές που ε, έχουν ήδη υπογραφεί και ε, να κάνουμε μια αξιολόγηση εκεί και να δούμε αν τηρούνται όλες οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι συμφωνίες που υπογράφονται είναι αποτελεσματικές για το στόχο που προσπαθούν να επιτύχουν. Και τέλος, Όσον αφορά την Κίνα, πέραν ε, όλων των προβλημάτων που είναι γνωστά της πάση για το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς και τη μη εφαρμογή της παρούσας μεθοδολογίας, εμένα με ανησυχεί και κάτι ακόμα. Πολλά κινέζικα προϊόντα φτάνουν από τα λιμάνια μας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να πληρούν την νομοθεσία και τις απαιτήσει που υπάρχουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να ελέγχονται όλα όσα εισέρχονται και υπάρχουν και διαφορετικά κριτήρια σε κάθε λιμάνι, όλα αυτά έρχονται να πλήξουν την ε, βιομηχανία μας. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει συνεργασία μεταξύ εμπορίου και τελωνίων, ώστε να υπάρχει καλύτερη εναρμόνιση και έλεγχη, ώστε πραγματικά αυτά τα οποία φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρούν τις ε, προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές. Ευχαριστώ. Η κυρία Μόσκα. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να συγχαρώ την Επίτροπο για τη ε, δραστηριότητες της ε, στα εμπορικά ζητήματα και τις επιτυχίες που επέτυχε στη διάρκεια αυτού του έτους. Δύο θέματα. Πρώτον, η Κίνα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Ξέρουμε ότι εχθές ε, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση, επομένως θα χρειαστεί και λίγος χρόνος για να τα επεξεργαστείτε όλα τα στοιχεία. Αλλά υπάρχουν πιέσεις και συζητήσεις και πέραν των διαβουλεύσεων έγιναν και από εξωτερικές πλευρές και στα θεσμικά όργανα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πολιτική μας ομάδα εκφράστηκε επί του ζητήματος. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κατά πόσον θα γίνουν σεβαστά. Δεν ξέρω, δεν ε, άκουσα ίσως αυτό το σημείο της παρέμβασής σας. Θα γίνει σεβαστή η προθεσμία που είχε προβλεφθεί για να μας υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση τον Ιούλιο για το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα και σε ποιο επίπεδο λεπτομέρειας έχετε φτάσει και μετά από τα αποτελέσματα της ε, διαβούλευσης ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν αναφέρθηκε και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Πού βρισκόμαστε στη συζήτηση για τη συμφωνία για τα green goods, για τα πράσινα αγαθά. Υπήρχαν πολλές ελπίδες, αλλά φαίνεται ότι έχουν αντιμετωπιστεί κάποιες δυσκολίες και ελπίζω ε, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επίτροπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Χαίρομαι που δηλώσατε σαφώς ότι η Κίνα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί η οικονομία της αγοράς. Νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικό. Και νομίζω ότι πρέπει να επαγρυπνούμε, όπως είπατε και εσείς ε, πολύ καλά, να εξετάζουμε περιβαλλοντικά θέματα, θέματα εργατικού δικαίου και dumping που θα μπορεί να προκύψει με την Κίνα διότι επηρεάζει την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη στη σιδηρουργία, στη, στα κεραμικά κλπ. Το θέμα των λιμένων είναι πολύ σημαντικό. Εγώ επισκέφτηκα το λιμάνι της Γένοβας, ήταν και συνάδελφος Μπεγκίν μαζί μου, και εκεί μα είπαν ότι το θέμα των τελωνίων είναι τελείω διαφορετικό από το ένα ευρωπαϊκό λιμάνι στο άλλο και πράγματα τα οποία επιτρέπονται σε ένα λιμάνι μπορεί να μην επιτρέπονται σε κάποιο άλλο. επομένω υπάρχει σοβαρή στρέβλωση. Επίση, να επαναλάβω αυτά που είπε και η Μακουλάδα για τα θέματα τη Λατινική Αμερική, το θέμα του σημερινού το σχολιάσουμε. Γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια του Συμβουλίου, αλλά ε, με την πτώση τη τιμή του πετρολαίου, με το σεισμό, είναι, θα είναι πάρα πολύ σοβαρό να μείνει το Εκουαδόρ χωρίς την προτιμησιακή συμφωνία που διαθέτει αυτή τη στιγμή και να πρέπει να καταβάλει δασμούς από 1η πρώτου του 2017. Αυτό μπορεί να πλήξει πολύ σοβαρά τη χώρα και αυτούς, αλλά και την Ευρώπη πιστεύω. Το θέμα του Μεξικού αναφέρθηκε επίσης, ε, να ξέρουμε τι γίνεται με τον εξυγχρονισμό της συμφωνίας και η κατάσταση στο Μερκοσούρ. Νομίζω ότι υπάρχει μια ευκαιρία με την ε, Προεδρία του Μάκρη που είπε ότι είναι διατεθειμένος να ξαναξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, αλλά υπάρχει και το θέμα της αστάθειας στη Βραζιλία. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό θα επηρεάσει τις συζητήσεις με το Μερκοσούρ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ κύριε Σούστερ, ευχαριστώ κύριε Μάμστρομ. Να ασχοληθώ με δύο θέματα που είναι για μένα σημαντικά Είπατε ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την εφαρμογή των συμφωνιών και την παρακολούθησή τους, καταλαβαίνω. Αλλά τι θα πρέπει να γίνει, ποιες δομές πρέπει να αλλάξετε, ποιες πιστώσεις πρέπει να προβλέψετε για να γίνει αυτό. Χρειάζεται να υπάρχει επαρκές προσωπικό στην Κομισιόν. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να εφαρμοστούν πλήρως οι φιλόδοξες προβλέψεις των συμφωνιών, τότε πρέπει να ασχοληθούν με το θέμα αυτό διάφορες γενικές διευθύνσεις. Για παράδειγμα, η συμφωνία με την Αφρική και την Καραβική ε, για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αν είναι όντως βιώσιμη η στρατηγική μας ε, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική ε, συνεκτική. Τι θα γίνει γι' αυτό. Υπάρχουν σκέψεις για το πώς θα οργανώσετε αυτή την παρακολούθηση γιατί επειδή έχει τόσο φιλόδοξες διατάξεις ε, η συμφωνία αυτή, πρέπει να διαπιστώσουμε ε, εάν όχι απλώς υπογράφονται, αλλά και αν εφαρμόζονται. Πρέπει να έχουμε συνολικά λοιπόν μια συνεπή πολιτική. Δεύτερον, συμφωνίες ε, εταιρικής σχέσης με τους γείτονές μας στην Ανατολική Ευρώπη. Με εξέπληξε το ότι θα υποβληθεί πρόταση απελευθέρωσης θεωρήσεων με την Ουκρανία χωρίς να αναφερθούμε καθόλου στην ε, Ολλανδία και τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Είδαμε ότι εκεί κατά πλειοψηφία οι Ολλανδοί απέρριψαν αυτή τη συμφωνία. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις ε, πολιτικές ε, ελπίδες που είχαμε συνδέσει με τις συμφωνίες αυτές σύνδεσης ε, τελικά δεν ε, προχωράνε. Ε, αναφέρθηκε ο κύριος Σόλτ στην Μολδαβία. Πείτε μας εσείς πώς το βλέπετε και πώς θα προχωρήσουν οι σχέσεις μας με την Ρωσία. Διότι οι χώρες αυτές συνορεύουν με τη Ρωσία και από ό,τι είχα καταλάβει μέχρι πρόσφατα είχε συνδεθεί η στάση που θα είχαμε έναντι των χωρών αυτών με τη στάση μας έναντι της Ρωσίας. Τι θα κάνουμε λοιπόν, υπάρχει προσπάθεια αναθεώρησης της ε, αντιμετώπισης αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η ε, Άγνες. Συγγνώμη, αλλά πατούσα λάθος κουμπί. Σας συγχαίρω για τις φιλοδοξίες σας. Ε, Ω προ το θεματολόγιο και τι πρωτοβουλίε που έχετε θέσει για την εμπορική πολιτική, δεν νομίζω ότι θα είμαι η τελευταία που σα επενεί. Θα ήθελα όμως ε, παρόλα αυτά να το κάνω. Δεύτερον, οι συνάδελφοι έχουν θέσει πολύ ε, ενδιαφέροντα ερωτήματα ήδη. Θα είμαι πολύ σύντομη λοιπόν. Υπάρχουν και άλλες φήμες, πέρα από αυτές που ανέφερε η Μαρίκα, Κυκλοφορεί μια φήμη βάσει της οποίας επειδή δεν θέλουν οι Αμερικανοί να χορηγηθεί το καθεστώς οικονομίας αγοράς ε, στην Κίνα, μας απειλούν ότι αν το κάνουμε αυτό θα σημάνει και το τέλος των διαπραγματεύσεων TTIP. Κυκλοφορούν πάρα πολλές φήμες για αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα ή δυνατόν να τις διαψεύσετε ή να τις επιβεβαιώσετε αυτές τις φήμες. Είμαι από την Ολλανδία, όπως ξέρετε, και όπως και ο συνάδελφος Σούστερ, ανησυχώ κι εγώ για το μέλλον ε, των εμπορικών συμφωνιών υπό το φως ε, των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος στην Ολλανδία. Γίνεται συλλογή υπογραφών ήδη για το επόμενο δημοψήφισμα για τη ΣΥΤΑ αυτή τη φορά. Έχετε προβλέψει κάτι σχετικό. μήπως ε, γίνει σαφέστατα η διάκριση ανάμεσα στο εμπορικό κομμάτι αφενός και αφετέρου ρίδρες περί προστασίας των επενδύσεων και κανονιστικών ρυθμίσεων. Αφετέρου, μήπως δεν πρέπει να είναι μεικτή η συμφωνία. Ε, μεικτής αρμοδιότητας δηλαδή, μήπως πρέπει να είναι αποκλειστική ενωσιακής αρμοδιότητας. Και τι προβλέπετε για τη Σιγκαπούρη, για την ε, απόφαση του δικαστηρίου, διότι ε, και γι' αυτό, γι' αυτή τη σύμφωνα εξετάζουμε το θέμα της αποκλειστικής ημεικτή αρμοδιότητας. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν μας δίνατε απαντήσεις για αυτά τα ζητήματα. Η κυρία Ρένα, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, διότι ως επιτοπλίστων τα έτσαν τα ερωτήματα οι συνάδελφοι για τη Σύμβαση Μαυρικίου, για την διαμεσολάβηση. Έχουν γραφτεί πολλά ε, για αυτό το ζήτημα και η Γενική Συνέλευση του ΙΕ το 2014 επικύρωσε μια σύμβαση βάσει της οποίας ε, υπάρχει δυνατότητα μηχανισμού διαφάνειας ανάμεσα σε αυτές τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί όμως πριν το 2014 ήδη. Και φαίνεται ότι έχει ε, μπλοκαριστεί διαδικασία σε επίπεδο κρατών μελών. Ε, ε, γιατί, τι έχει γίνει, δεν ε, υπάρχει βούληση να επικρατήσει διαφάνεια για το ISDS, για τη το μηχανισμό διευθέτησης δηλαδή των, των διαφορών για τις επενδύσεις ή αμφισβητείται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα των επενδύσεων θεωρούν, δηλαδή την εθνική αρμοδιότητα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε Ζήκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι τα καθήκοντά σας και τα δικά μας τα καθήκοντα, το να είμαστε ρυθμιστές δηλαδή για την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα είναι ε, σημαντικός ε, πολύ περισσότερο λόγω της κατάστασης που βιώνει η Ευρώπη, της κρίσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, του γεγονότος ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους. Και νομίζω ότι η εμπορική πολιτική, καθώς και όλα τα υπόλοιπα τα οποία δεν θα αναφέρω γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά, ε, είναι πολύ σημαντικά και για να ανακτηθεί εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό λοιπόν το οποίο κρατώ εγώ είναι ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Για τα μεγάλα ζητήματα τα οποία συζητούμε, ε, δεν θα επαναλάβω τα της Κίνας, ε, την TTIP και τις άλλες εμπορικές συμφωνίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ε, τα αντιμετωπίσουμε σωστά και να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Δεν μπορούμε να έχουμε ψευδεστήσεις και να σιωπιούμε. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας γιατί πρέπει να δώσουμε απαντήσεις, διότι οι απαντήσεις περιμένουν χώρες όπως η δική μου, η Ιταλία, όπου το βιομηχανικό σύστημα είναι ε, πιεσμένο και ξέρουν τι συνέπειες μπορεί να έχει αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς της Κίνας και επομένω, ε, ξέρουμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο να βρούμε την καλύτερη λύση. Όπως επίσης και η TTIP για τι γεωγραφικές ενδείξεις που μας αφορούν εμά που βρίσκονται σε, στην πρώτη γραμμή σε σχέση ε, με τα θέματα που συζητάμε σήμερα στην ΙΜΚΟ και που πέρασαν με την ψηφοφορία και θα πάει στην ε, Ολομέλεια. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που είπε ο συντονιστή μα, ο κύριος Κάσπαρη. Επίση, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας πω ότι κατά την άποψή μου είναι πολύ επιθετική η εμπορική πολιτική μας όταν ξεκινάει η συνεργασία μας με τις τρίτες χώρες, κυρίως σε σχέση με την Νότια Ευρώπη και κυρίως το νότο της Ιταλίας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δίνουμε τόσα πολλά από πλευράς οικονομικής στήριξης. Εγώ είμαι εισηγητής για την Τινησία ε, και θα δοθούν 500 εκατομμύρια ευρώ, εκεί ε, κάνουμε πιο ήπιες τις διαδικασίες, αποφασίζουμε να μην υποβάλουμε τροπολογίες και όλα αυτά, εντάξει, αλλά προσοχή, ε, υπάρχει εμπορική πτυχή όπου τα πορτοκάλια, το ελαιόλαδο, το ο όλα αυτά καταπατούνται και οι γεωγραφικές ενδείξεις επίσης. Επομένως, δεν είναι μόνο εμπορική ζημία, υπάρχει και ζημία ως προς την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά την ε, εκπόνηση αυτής της πολιτικής. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε γιατί νομίζω ότι θα αυξηθεί η έλλειψη εμπιστοσύνη των πολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σμουέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε σήμερα. Εγώ βλέπω ένα παράδοξο σε όλα αυτά. Ε, διαδοχικά σας επενούν οι συνάδελφοι, βλέπουν ότι σημειώνεται πρόοδος, ε, όλα βαίνουν αισίως, ε, όντως σε σχέση με τον προκάτοχό σας. Όμως ταυτόχρονα ε, στην Ευρώπη επικρατεί ένα κλίμα ε, απογοήτευσης, ε, κυρίως για αυτές τις συμφωνίες. δεν μιλάω μόνο για την TTIP, η συμφωνία με την Ουκρανία, σε αυτή την ε, φιλοευρωπαϊκή χώρα ήταν αρνητικό, αρνητική έκβαση του δημοψηφίσματος. Δεν πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί, διότι ε, υπάρχει μια επανάσταση που πρέπει να γίνει ως προς την μεθοδολογία, ως προ την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις αυτών των συμφωνιών. Αυτό είναι απαραίτητο για μας, ε, διότι όποιον και να ρωτήσετε, όποιο πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απορρίψει αυτά που κάνατε, διότι είναι Ελάχιστη διαφάνεια. Ναι, λέτε ότι έχει σημειωθεί πρόοδο. Βέβαια, όταν ξεκινάμε από τον πάτο, μόνο καλύτερα μπορεί να πάει. Και ε, δεύτερον, υπερασπίζεστε κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Και τρίτον, χρειάζεται χρόνο. Και επίση αυτή η διγλωσία πρέπει να σταματήσει. Λέτε, ναι, ναι, ναι, είμαστε φιλόδοξοι για να λαμβάνουμε δέσμευση. Όρια για τη ΣΕΤΑ, λοιπόν, χρειαζόμαστε ξεκάθαρη απάντηση. Ε, θα εφαρμοστεί προ, ε, προσωρινά ναι ή όχι. Για την ΤΤΙΠ θέλουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Μα, συγγνώμη, δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσει ω προ αυτά που ζητούμε για την TTIP. Κυκλοφορούν, οργιάζουν οι φήμε όμως ε, για το αντίθετο. Για την έγκριση των συμφωνιών από πλευρά ε, Κοινοβουλίου ε, λέτε ναι, αλλά λέμε, λέτε ότι δεν τελικά στην έκθεση αναφέρεται ότι δεν γίνεται να ενισχυθούν οι αρμοδιότητε του Κοινοβουλίου σε αυτό το τομέα. Και τέλος, ιδιαίτερα για τη Γαλλία, αλλά και για άλλε ευρωπαϊκέ ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε τι διαπραγματεύσει με το Μερκόσουρ και φαίνεται ότι διαπραγματεύεται τώρα με συμφωνία ε, που θα συμπεριλαμβάνει και το βόηο Κρέα. Πολλοί εκτροφή ε, θα ε, περιέλθουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και θα ενισχυθεί η τωρινή κρίση και το ξέρετε. Ευχαριστούμε. Κύριο Στάκουλ. Ευχαριστώ. Καλύτερα να βάλετε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Θα επανέλθω, πρέπει να φύγω για λίγο, θα επανέλθω. Τέλο πάντων, βάλτε τα ακουστικά και θα μιλήσω φιλανδικά για να ε, μιλήσω πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται την ΤΙΖΑ και τη ΣΕΤΑ και ξέρουμε ότι είναι πολύ διαφορετικές ε, αυτές οι συμφωνίες Υπάρχουν ε, ε, πολλά ε, περίπλοκα τεχνικά στοιχεία μέσα στις συμφωνίες. Τι γίνεται λοιπόν όταν υπάρχει επικάλυψη. Τι γίνεται όταν υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων και με ποιο τρόπο μπορείτε να επιτύχετε μια καλύτερη έκβαση στις διαπραγματεύσεις. Εντάξει. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπούχνερ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ασχοληθήκατε πρώτα απ' όλα με το δίκαιο εμπόριο. Γιατί εδώ χρειάζονται πολλές βελτιώσεις. Ε, πρέπει να σας πω ότι με απαγοήτευσαν τα αποτελέσματα της διάσκεψης στο Ναϊρόμπι γιατί δεν επέλυσε τα πραγματικά προβλήματα. Όπως προηγουμένως έχουμε το πρόβλημα ότι στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες δίνουμε τρομερές επιδοτήσεις στα γεωργικά προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά κατόπιν τα πετάμε στις αγορές των αναπτυσσομένων χωρών και κατά συνέπεια καταστρέφουμε τη δική τους γεωργία. Φέρουμε λοιπόν και εμείς την ευθύνη για πολλά προβλήματα σε αυτές τις χώρες. Είμαστε συνυπεύθυνοι. Οπότε η ερώτηση αλλά και παράκλησή μου. Σας παρακαλώ να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Τι θέλετε να κάνετε για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε. Να πω όμως και εγώ κάτι για το αίτημα των κυρίων Τζίκο και Μορέλ. Έχουμε τη συζήτηση αυτή τη στιγμή για την εμπορική πολιτική της Ένωσης. Λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει δυσπιστία προς τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Δεν θα έπρεπε βασικό στοιχείο του επόμενου προγράμματος εργασίας σας να είναι πώς θα επανέλθει η εμπιστοσύνη στην εμπορική πολιτική. Να μην προσπαθήσετε να κάνετε τόσο πολλά επιμέρους, αλλά να προσπαθήσετε να ανακτήσετε την εμπιστοσύνη της κοινή γνώμης για την εμπορική πολιτική. Γιατί αλλιώ, ό,τι και να αποφασίσουμε εδώ πέρα, ό,τι θαυμάσια και να αποφασίσουμε, δεν θα έχουμε μαζί μας ένα μεγάλο τμήμα της κοινή γνώμης. Η κυρία Μάλστρομ. Να ξεκινήσω με αυτό. Καταρχάς ευχαριστώ όλους τους ευρωβουλευτές για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα που θέσατε. Βεβαίω υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη όχι μόνο τη εμπορική πολιτική, αλλά γενικότερα έναντι τη πολιτική στην κοινή γνώμη διαφόρων χωρών. Και υπάρχουν κάποιε πολιτικέ δυνάμει που εκμεταλλεύονται αυτή την ε, έλλειψη εμπιστοσύνη και υπονομεύουν τι προσπάθειέ μα και διασπείρουν φήμε, πολλέ εκ των οποίων είναι εντελώ αβάσιμε. Αυτό που θέλησα να σας πω και τώρα και την προηγούμενη φορά είναι ότι ναι, αλλάξαμε, προσαρμόσαμε την εμπορική μας πολιτική, είναι πολύ πιο διαφανής. Ποτέ στο παρελθόν η εμπορική πολιτική της Ένωσης δεν, είναι, δεν ήταν τόσο διαφανής όσο σήμερα. Ξέρω ότι δεν θεωρείται ότι είναι επαρκώς διαφανής, αλλά βήμα το βήμα καθίσταται πιο διαφανής δημοσιεύουμε τις διαπραγματευτικές εντολές, ε, την τεκμηρίωση, συζητούμε με τα κράτη-μέλη, δεσμευόμεθα να το κάνουμε, ορισμένες, ε, ορισμένα κράτη-μέλη αντιστέκονται περισσότερο, αλλά και με τους εταίρους μας. Κάθε φορά πριν ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις λέμε ναι, ναι, δεσμευόμεθα να υπάρξει διαφάνεια. Και ε, ακούσαμε και τη γνώμη πολλών χωρών. Ε, όπου τους ε, λέμε ότι είναι καλό να ανοίξουν τις αγορές τους γιατί έτσι θα δημιουργήσουν και ευκαιρίες και θέσεις εργασίας για όλους. Αλλά η εμπορική πολιτική δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, είναι θέμα επίσης να υπάρξει διάδοση των αρχών για τις εργατικές ε, προδιαγραφές, για τη βιωσιμότητα και να υπάρξει δέσμευση, δέσμευση για αυτά με την κοινωνία των πολιτών, με τα συνδικάτα της ΜΚΑΟ, τις επιχειρήσεις, την κοινή γνώμη με έναν εντελώ πρωτοφανή τρόπο ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εμπορικής μας πολιτικής. Και εστιάζουμε και στην εφαρμογή των συμφωνιών. Να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή όντω θα είναι συνεπής με το περιεχόμενο των συμφωνιών και εάν διαπιστώσει η κοινή γνώμη ότι υπάρχει μέσω της εμπορικής πολιτικής περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη απασχόληση και εδώ και στους εταίρους μας και ότι προωθούμε σημαντικές αξίες και ότι όντως αλλάζει τα πράγματα, τότε νομίζω ότι σταδιακά θα επανέλθει η εμπιστοσύνη. Αλλά αυτό δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Και η Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί και το κάνουμε. Και οι εργαζόμενοι στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου ε, εργάζονται σκληρά, κάνουν καταπληκτικά πράγματα με περιορισμένου πόρου. Ενώ οι απαιτήσει αυξάνονται καθημερινά, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μα. Πρέπει να δεσμευτούν και τα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ να ξεκινήσω καμία εμπορική διαπραγμάτευση χωρί εντολή από τα κράτη-μέλη. Το ξέρετε αυτό. Και συμμετέχετε κι εσεί σε αυτή τη διαδικασία. Τα κράτη-μέλη λοιπόν πρέπει να δεσμευτούν. Και όταν βγαίνουν και επικρίνουν την Κομισιόν, το καταλαβαίνω. Εντάξει, βεβαίω. Ε, δουλειά μα είναι να μα επικρίνουν. Αλλά δεν μπορούμε εμεί να πουλήσουμε, να πωλήσουμε, να παρουσιάσουμε την εμπορική πολιτική ε, έρχονται στι διαπραγματεύσει και λένε ξεκινήστε διαπραγματεύσει, ε, κάντε το πιο γρήγορα, πάτε TTIP. Και μετά πάνε πίσω στη χώρα του και λένε όχι, όχι, δεν θα πρέπει να διαπραγματευτούμε αυτή τη χώρα. Δεν καλό το TTIP. Ειλικρινά πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια, μια σοβαρότητα. Κάποιοι εθνικοί ηγέτε πρέπει να το κάνουν. Εμεί έχουμε αλλάξει σε σημαντικό βαθμό την εμπορική πολιτική και ελπίζω ότι σταδιακά θα παρέλθει η εμπιστοσύνη, αλλά δεν αρκεί η δική μα ε, δράση. Πρέπει να μα στηρίξετε κι εσεί για τι ερωτήσεις σας. Κύριε Γκασπάρη, έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως, ε, παλεύουμε για να βγάλουμε ε, κάποιες προτάσεις. Για τα ορυκτά από ε, εμπόλεμε ζώνες, ναι, θα υποβάλουμε προτάσεις. Θα προχωρήσει ο τριμερής διάλογος. Ελπίζω να καταλήξει πριν τις διακοπές. Για το IPI. Για τα θέματα πνευματικής διοκτησίας θα επιταχύνουμε. Ελπίζουμε, Προεδρία, να το θέσει στην ημερήσια διάταξη. Γιατί πρέπει να προωθηθεί το θέμα αυτό, γιατί οι πολίτες ε, περιμένουν αποτελέσματα. Και θέλουμε να έχουμε και σωστά μέσα ε, άμυνας ε, στον εμπορικό τομέα, που δεν πρέπει φυσικά ε, να το χρησιμοποιούμε υπερβολικά, αλλά πρέπει να τα εφαρμόζουμε όταν υπάρχουν θέματα ε, αθέμητο ανταγωνισμού και στο θέμα της Κίνας και για τη χαλιβουργία υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε νομικά ε, στέρεα μέσα για την καταπολέμηση των βασανιστήριων. Έχουν γίνει ορισμένα και δεν είμαι σίγουρη αν θα τα καταφέρουμε κατά την Ολλανδική Προεδρία. Και για τη διπλή χρήση βεβαίως λυπάμαι που έχουμε καθυστερήσει. Είναι πολύ περιπλοκό θέμα αλλά ελπίζω να μπορέσουμε μετά τις διακοπές να σας υποβάλουμε πρόταση. Το παλεύουμε. Σιγκαπούρη. Δεν ξέρουμε πότε το, το δικαστήριο θα διακρινίσει την κατάσταση για τις μικτές συμφωνίες. Ε, ελπίζω το φθινόπωρο και την περιμένουμε με ανυπομονησία, αλλά δεν, δεν ξέρω. Δεν έχω πληροφορίες γιατί δεν υπάρχουν διαρροές από το δικαστήριο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ βέβαια είναι καλές οι συζητήσεις με τη Σιγκαπούρη. Κάποια αντιπροσωπεία πήγε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Ε, πολλά έχουν κλείσει, αλλά συζητούμε για το θέμα του κεφαλαίου για τις επενδύσεις και ελπίζω να προχωρήσει. Ούτω ώστε όταν θα έχουμε τη διευκρίνηση από το δικαστήριο να περάσουμε σύντομα στη φάση εφαρμογής. Κύριε Μάρτιν, και εσείς αναφερθήκατε στα μέσα εμπορικής άμυνας και τη διπλή χρήση, ναι, οπότε απάντησα, για την Ταϊουάν. Πρόσφατα έγιναν εκλογές, ξέρετε. Και η κυβέρνηση θα αναλάβει καθήκοντα στις 20 Μαΐου. Οπότε μετά θα ξεκινήσουμε διερευνητικέ επαφές. Όταν αναλάβει. Για την Ινδία. Δυστυχώς δεν έχουμε προχωρήσει πολύ. Έχουμε κάνει πολύ διαφορετικές προτάσεις από ομάδες εργασίας για επιτάχυνση, αλλά δεν ήταν σε θέση να τις αποδεχθούν όταν συναντηθήκαμε. Έστειλαν ένα ε, πολύ ειλικρινές ε, γράμμα όπου περιγράφονται τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης κορυφής. Δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικά, αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να συζητήσουμε. Θα έχουμε διάφορες ευκαιρίες, ο ΣΑ, 20 οποτεδήποτε συναντώμεθα με τον Υπουργό Εμπορίου θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο. Για το νομικό έλεγχο και τη μετάφραση, ναι, συμφωνώ. Έχουμε 23 γλώσσες και είμαστε δεσμευμένοι από τον νόμο να έχουμε τις μεταφράσεις. Προσπαθούμε να επιταχύνουμε το νομικό έλεγχο. Είμαστε σε επαφή με την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου για να μην κάνουμε δύο φορέ την ίδια δουλειά. Νομίζω ότι αν συνεργαστούμε καλύτερα μεταξύ των σχετικών υπηρεσιών Επιτροπής και Συμβουλίου μπορούμε να επιταχύνουμε. Ίσως ε, να κρατήσει μόνο ένα τρίμηνο, αλλά πρέπει να γίνει αυτός ο έλεγχος. Δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε. Οπότε έρχομαι στις ε, ερωτήσεις για το προσωπικό. Τα κράτη-μέλη και εσείς και διάφοροι άλλοι και εμείς οι ίδιοι ε, αναλαμβάνουμε νέα καθήκοντα και εσείς μας αναθέτετε νέα καθήκοντα. Αλλά όλα αυτά σημαίνει προσωπικό και το προσωπικό μας δουλεύει πολύ σκληρά. Αλλά έχουμε δουλειά και για εκατοντάδες άλλους, αν τους είχαμε. Αν πρόκειται να κάνουμε όλα αυτά που μας ζητάτε, διαφάνεια και τα μέσα άμυνας. Γιατί δεν δουλεύετε όπως ε, οι Αμερικανοί τόσο γρήγορα. Αλλά αυτοί έχουν εκατοντάδες άτομα που ασχολούνται με το θέμα αυτό, ενώ εμείς όχι. Υπάρχουν πολλές φήμες για το ανώβερο. Ε, ο, κύριε, ο πρόεδρος Ομπάμα θα είναι εκεί, εγώ θα είμαι εκεί, διάφορα άλλοι επίτροποι, πρέσβεις. Θα υπάρξουν εκδηλώσεις ε, μια εβδομάδα. Ε, θα οργανώσει η καγκελάριος Μέρκελ ένα δείπνο όπου θα συμμετάσχουν πολλοί. Και ελπίζω ότι θα γίνει και μια συζήτηση για το TTIP. Τώρα τι θα προκύψει δεν ξέρω. Αλλά προχωράμε για το TTIP. Κάθε εβδομάδα σχεδόν ε, γίνονται συναντήσεις. Αλλά πολλά θέματα ακόμη πρέπει να συζητήσουμε. Και εμείς και οι Αμερικανοί έχουμε πει σαφώ ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ένα ε, TTIP ε, light, ένα TTIP πολύ περιορισμένο. Το θέμα δεν είναι να περιορίσουμε κάποιου δασμού. Δεν θα ήταν αυτό αποτέλεσμα για όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει. Πρέπει να προχωρήσουμε για τι κρατικέ προμήθειε, για τι υπηρεσίε, του γεωγραφικού δείκτε που ανέφερε, ανέφερε ο κύριο Ζήκου και άλλοι. Έχει σημειωθεί ουσιώδη πρόοδο στον κανονιστικό τομέα. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε κάποιο απολογισμό κάποια στιγμή για να κάνουμε κάποια θετική δήλωση για τη σημασία του TTIP, αλλά θα δούμε την Παρασκευή ή Δευτέρα. Απαντώντας τον κύριο Σόλτς, ναι, θέλουμε να υπάρχει δίκαιο εμπόριο, προγράμματα και πρακτικές δικαίου εμπορίου, θέλουμε να τα βοηθήσουμε και να καθορίσουμε ευρωπαϊκές παραμέτρους για το τι σημαίνει αυτό και προσπαθούμε επίσης να εφαρμόσουμε την πρόταση που κάνετε και εσείς και ο κύριος Μάρτιν για αυτά τα βραβεία για τις τοπικές πρωτοβουλίες δικαίου εμπορίου. Ελπίζω και αυτό να προχωρήσει. Για τον ΠΟΕ. Κάνουμε εμπεριστατωμένες συζητήσεις για να προχωρήσουμε. Μέχρι το φθινόπωρο θα θέλαμε να δούμε τι θα επιτύχουμε ε, στη συνάντηση MC11 που θα είναι η επόμενη συνάντηση τον Σεπτέμβριο του 2017. Οι φίλοι του ΠΟΕ, και είναι πολλοί σε διάφορες περιοχές του κόσμου, θέλουν να πιέσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να διατυπώσουμε ένα ρεαλιστικό αλλά και φιλόδοξο θεματολόγιο Γενικά το συζητάμε αυτό συνέχεια με τα κράτη-μέλη. Γίνεται διάλογος και θα οργανωθεί την ερχόμενη Τρίτη και ένας διάλογος της κοινωνίας των πολιτών. Θα συζητήσουμε και, στο, και στη Σανγκάη και στο Παρίσι το μέλλον του ΠΟΕ. Σιγά σιγά λοιπόν προχωράμε. Και φυσικά η συμβολή σας είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Α, το, τις απώλειες πόρων από τους δασμούς βεβαίως, το λαμβάνουμε υπόψη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε όλες μας, ε, όλοι μας οι κανόνες να γίνονται σεβαστοί σε όλα τα λιμάνια, από όλα τα τελωνία. Να δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Και επανέρχομαι στο θέμα της απώλειας ε, από τους δασμούς. Θα υπάρξει αυτόματη ε, αντικατάσταση από το ύψος του ΑΕΠ που συμβάλλουν τα κράτη-μέλη. Όπως ξέρετε κάνουμε διαπραγματεύσεις με την Κίνα, όπως συζητάμε μερικά αυτά τα θέματα για να υπάρξει πιο θεμητός ανταγωνισμός, περισσότερη διαφάνεια στις σχέσεις μας στον τομέα των επενδύσεων με την Κίνα κυρία Κέρτσον Ντάλινγκ. Ναι, έχω ακούσει και εγώ ότι υπάρχει δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίκειται. Βεβαίως δεν θέλουμε να παρέμβουμε ως Κομισιόν. Αλλά βεβαίως ε, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική διατυπώνεται από την Κομισιόν μετά από την συμβολή του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών και καμία εμπορική συμφωνία δεν συζητείται χωρίς ε, ομόφωνη εντολή από τα κράτη-μέλη και συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε βήμα που κάνουμε σε κάθε διαπραγμάτευση ελέγχουμε και πριν και μετά και με εσά και με τα κράτη-μέλη. Υπάρχει αυτή η συνεχής παρακολούθηση. Έχετε ειδικέ ομάδες εργασίας για κάποιες από τις διαπραγματεύσεις και φυσικά και η ίντα τις παρακολουθεί και μέσω της πρωτοβουλίας Εμπόριο για Όλους κάνω ό,τι μπορώ ούτω ώστε όλες οι διαπραγματεύσεις που κάνουμε να έχουν το ίδιο επίμενο διαφάνειας με το TTIP. Δημοσιεύουμε τις εντολές, την τεκμηρίωση, κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε η γνώμη έξω από την απομόνωση μόνος στις Βρυξέλλες να ενημερώνονται. Έχω υποσχεθεί όχι σε εσά εδώ αλλά στο Κοινοβούλιο ότι αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για κάποια εμπορική συμφωνία, δεν θα υπάρξει προσωρινή εφαρμογή μέχρι να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, ούτε το TTIP, ούτε καμία άλλη συμφωνία δεν θα εφαρμοστεί προσωρινά πριν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Τώρα το θέμα για το μεικτό χαρακτήρα είναι άλλο, αλλά οι συνομοθέτες είναι τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Με συγχωρείτε, θέλετε να σχολιάσετε κάποιες αποφάσεις των κρατών μελών για το θέμα του μεικτού χαρακτήρα. Γιατί αν εφαρμόζεται προσωρινά ήδη η συμφωνία, Ε, γιατί αυτό καταλάβαμε από κάποιον εκπρόσωπο της Επιτροπής για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας για την Ουκρανία. Όπως ξέρετε η χώρα μου καταψήφισε αυτή τη συμφωνία. Δεν θέλω να είμαστε σε μια τέτοια ασαφή κατάσταση. Η κυρία Μάλστρομ. Εάν είναι μεικτή ή όχι μια συμφωνία, η Κομισιόν κάνει μια πρόταση από αυτού και κατόπιν αποφασίζουν τα κράτη-μέλη και πάντα αποφασίζουν ότι είναι μεικτή. Γι' αυτό νομίζω ότι και η Επιτροπή και το Συμβούλιο και πολλοί άλλοι αναμένουν τη γνώμη του δικαστηρίου. Γιατί η συνθήκη τη Λισαβόνα ε, ήταν ένα βήμα προ τα μπρο, ούτω ώστε η Ένωση από πλευρά των κρατών μελών και των εκλεγμένων εκπροσώπων του να μπορεί να κάνει εμπορικέ συμφωνίε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, αλλά αυτό λέει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Αλλά τώρα η ερμηνεία ε, περιέχει κάποιε ασάφειε και ελπίζω ε, το δικαστήριο να μα δώσει κάποιε καταυντήρε γραμμέ. Αλλά όπω ξέρετε, το δημοψήφισμα ε, αφορούσε συνολικά τη Συμφωνία Σύνδεσης και η απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι εκτός των Συμφωνιών ε, Σύνδεσης, κύριε Σόλτς. Περιμένουμε η Ολλανδική κυβέρνηση να μας δώσει κάποιες ενδείξεις για το πώς ε, ερμηνεύουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και τι θέλουν να κάνουμε περαιτέρω. Περιμένουμε. Αλλά ό,τι και αν προκύψει για το μεικτό χαρακτήρα από την απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να το συζητήσουμε για να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Και εάν κάθε εμπορική συμφωνία τώρα θα υπόκειται σε συνολικά ή επιμέρους δημοψηφίσματα, ε, τότε είναι ζόρικα τα πράγματα. Πρέπει να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι κυβερνήσεις εκπροσωπούν το λαό. Και εσείς εκπροσωπείτε το λαό. Τώρα δεν πρόκειται εγώ να κάνω αποτίμηση του ποιος είναι πιο δημοκράτης. Για το Μερκοσούρ και τη Βραζιλία, η Μακουλάδα. Ναι, πράγματι υπάρχουν κάποιες ε, αναταράξεις, να το πω, στη Βραζιλία. Η Ουρουγουάια έχει αυτή τη στιγμή την Προεδρία του Μερκοσούρ και θα συνεχίσουν να ασχολούνται με το θέμα του εμπορίου ακόμα και όταν η Προεδρία μεταβιβαστεί στη Βενεζουέλα γιατί δεν συμμετέχουν στο εμπορικό κομμάτι αυτή. Ε, επομένως, ε, εμεί ασχολούμαστε με την Ουρουγουάη και μας έχουν δώσει σαφή ένδειξη ότι η Βραζιλία έχει δεσμευτεί επ' αυτού και μέχρι να πάρουμε άλλη ένδειξη πρέπει να του εμπιστευτούμε. Γνωρίζουμε την προθεσμία για τον Ισημερινό, το ανέφερε και ο κύριο Πίσα. Ε, εμείς κάναμε αυτό που μας αναλογεί και ελπίζω να βιαστείτε εσεί και το Συμβούλιο, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσει. Και νομίζω ότι Υπάρχει και το αίτημα αυτό, το έχουμε κάνει και έκκληση στο Συμβούλιο. γιατί τη Χιλή υπάρχουν προετοιμασίες για τον εξυγχρονισμό αυτής της συμφωνίας. Χρειαζόμαστε και εμείς όμως αυτή τη χρονιά για να κάνουμε προετοιμασία. Δεν θέλω να σας δώσω ημερομηνίε, αλλά μάλλον ε, για του χρόνου. Πρέπει να δούμε και τα θέματα της εφαρμογής. Το ρώτησε και ο κύριος ε, Σόλτς αυτό πρέπει να συνεργαστούμε. Μπορεί να βοηθήσουν τα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να συνεργαστούν οι διάφορε Γενικέ Διευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί συνεργαζόμαστε, λαμβάνουμε πολλά στοιχεία από τα κράτη-μέλη, από τι πρεσβείε, από την κοινωνία των πολιτών, από τον ίδιο τον κλάδο. Επομένω, προσπαθούμε να λάβουμε τις πληροφορίες για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ε, την κατάσταση της εφαρμογής και συμμετέχει όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό και αρχίζουμε να ε, εκπονούμε και μια πιο ευφυή στρατηγική για να το ελοπίσουμε. Κυρία Μόσκα, για τα πράσινα αγαθά. Ε, δυστυχώς ε, είναι στάσιμα τα πράγματα. Η Κίνα έχει κάποια προβλήματα τα οποία δεν έχουμε καταφέρει να επιλύσουμε μαζί τους ακόμα θα εκμεταλλευτούμε την ε, συνεδρίαση του ΟΣΑ στα τέλη Μαΐου-Ιουνίου για να συναντηθούμε με τον αρμόδιο για τα θέματα αυτά, να δούμε αν ε, μπορούμε να τα προχωρήσουμε, διότι οι συζητήσεις προχωρούν καλά κατά τα λοιπά, επομένως είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δείξουμε ότι η εμπορική ε, πολιτική μπορεί να συνεισφέρει και στους στόχους της COP21. Και αυτός είναι και ένας νέος τρόπος να εμπορευόμαστε, να διευκολύνουμε το εμπόριο σε πράσινα αγαθά, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν πολύ καλύτερα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Απάντησα για το Εκουαδόρ, το Μεξικό και το Μερκοσούρ, για την Κίνα και το χρονοδιάγραμμα, όπως σας είπα, πήγαμε πολλές απαντήσεις από τη δημόσια διαβούλευση, πρέπει να τα αξιολογήσουμε αυτά. Είναι σαφές ότι η Κίνα δεν είναι η οικονομία της αγοράς, εκπνέουν οι προθεσμίες ε, του πρωτοκόλου ε, προσχώρησης τους ε, και οι διατάξεις αυτές μας ενδιαφέρουν. Επομένως, ή η Κίνα θα φύγει από τον κατάλογο των χωρών που θεωρούνται οικονομία της αγοράς ή όχι και θα αλλάξει ο τρόπος που υπολογίζεται το, η καταπολέμηση του ντάμπινγκ. Και εάν αλλάξει και φύγουν από τον κατάλογο μπορούμε να προστατεύσουμε αυτά που έχουμε ήδη ή και για το μέλλον να έχουμε ισχυρούς μηχανισμούς εμπορικής άμυνας. Ε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Ε, πρέπει βέβαια να πάρουμε και τα στοιχεία από τη δημόσια διαβούλευση. Δεν μπορώ να σας δώσω τώρα χρονοδιάγραμμα, αλλά εάν κάνει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε σίγουρα χρειάζονται και χρόνο οι συνομοθέτες για να τα συζητήσουν. Η συζήτηση λοιπόν αυτή θα γίνει με τον Πρόεδρο και τη Γραμματεία. Αυτή τη στιγμή πλησιάζουμε και εμείς λίγο στο στόχο και πρέπει να αποφασίσει βέβαια και το Σώμα των Επιτρόπων. Δεν μπορώ να σας δώσω ακόμα ακριβή ημερομηνία γι' αυτό. Για την Ουκρανία απάντησα. Κυρία Γιόγκενης, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν πρέπει να αλλάξουν την νομοθεσία του για την ε, οικονομία τη αγορά τη Κίνα. Μόνο η Ευρώπη έχει νομοθεσία που προβλέπει ότι οι χώρε είναι είτε στον ένα κατάλογο ή στον όλο. Καμιά άλλη χώρα δεν έχει κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται λοιπόν νομική πρόταση. Μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που το υπολογίζουν σε ένα λεπτό. Δεν χρειάζεται να περάσει καν από το Κογκρέσο είναι λίγο πιο ελεύθεροι στην προσέγγιση τους δηλαδή. Σαφώς και συζητούμε με τους Αμερικανούς το θέμα και με πολλές άλλους από τους εταίρους μας. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μας απείλησαν ότι θα σταματήσουν τις διαπραγματεύσει στη TTIP αν εμείς κάνουμε κάτι τέτοιο, σας διαβεβαιώ. Για τα δημοψηφίσματα νομίζω σας απάντησα. Κυρία Αρένα, η σύμβαση που αναφέρεται μόνο η Πολωνία δεν την έχει υπογράψει και δεν το έχει κάνει για λόγους εθνικής αρμοδιότητας. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ευρώπη στο σύνολό της δεν έχει ε, υπογράψει, δεν έχουμε προσχωρήσει, λυπάμαι γι' αυτό. Κύριε Τσίκου, αναφερθήκατε σε πολλές από τις ευαισθησίες τις οποίες εξετάζουμε στην TTIP. Σίγουρα οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι ε, πολύ σημαντική προτεραιότητα. Νομίζω ότι γνωρίζετε ότι πιέζουμε να υπάρχει αντίστοιχο επίπεδο φιλοδοξία στην TTIP όπω έχουμε και στη ΣΥΤΑ. Οι Αμερικανοί έχουν τελείω διαφορετική παράδοση από αυτού και είναι πολύ περίεργο αυτό ο τρόπο για αυτού. Είναι λοιπόν λίγο παράδοξη αυτή η συζήτηση, αλλά αισιοδοξώ ότι θα βρούμε λύση. Ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Ιταλία και για πολλέ άλλε χώρε. Επίση, συνειδητοποιούμε ότι κάποια από τα προϊόντα ε, στον ε, πολιτιστικό τομέα είναι ευαίσθητα. Επομένως ε, και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη στις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, αλλά είναι αλήθεια ότι έχουμε και πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες για να ανοίξουμε αγορές για τα γεωργικά μας προϊόντα ε, στις χώρες του Μερκοσούρ, γαλακτοκομικά, για παράδειγμα, το να μην υπάρχουν δασμοί θα κάνει πιο ανταγωνιστική, τα, ανταγωνιστικά τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα. Κύριε Μορέλ, νομίζω ότι σας απάντησα στην αρχή την ερώτησή σας. Μπορεί να διαφωνείτε, αλλά πραγματικά προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τη μέθοδό μας. Ακούγονται πολλές φήμες, αλλά πολλές από αυτές είναι ψευδείς για την πρόταση για το Μερκοσούρ, για το Βόλιο Κρέα. Έχουμε προσαρμόσει την πρότασή μας σε σχέση με το 2004, αλλά δεν μπορούμε να απεμπολίσουμε εντελώ αυτά τα οποία είχαμε υποσχεθεί το 2004. Υπάρχουν κάποιες ποσοστώσεις, ε, θεωρώ ότι είναι λογικές. Σε αντάλλαγμα λαμβάνουμε πολλές άλλες δυνατότητες για το δικό μας ε, κλάδο του Βόλιου Κρέατος, αλλά και την κτηνοτροφία και τη Γεωργία Γέννη. Ο κ. Στάκουλα έφυγε για την αλληλοεπικάλυψη μεταξύ τίτη πτήσα. Ε, γιατί δεν έχουμε απάντηση. Θα γίνει υπουργική διάσκεψη για την Τίζα στις 21 Μαΐου, θα προεδρεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος εκεί, αλλά υπάρχουν ε, αρκετές χώρες αυτή την ομάδα, τελείως διαφορετικέ και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε καλύτερα στην TTIP για τις υπηρεσίες από ό,τι στην TISA. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Αν όχι, δεν το έκανα επίτηδες, κάποια μου διέφυγε ίσως. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ήσασταν πολύ ακριβείς και τηρήσατε και το χρόνο σας. Ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε επαφή. Ε, συνάδελφοι, μπορείτε να κάνετε προτάσεις στους συντονιστές οι οποίοι θα διαβιβάσουν το αίτημά σας στην διάσκεψη των Πρόεδρων. Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε σύντομα, υποθέτω, στο Ανόβερο. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Πρώτα απ' όλα, σημείο 15. Το πρωτόκολλο για τα προϊόντα καπνού. Είναι μόνο μία ψηφοφορία. Αλλά πριν ψηφίσουμε, να κάνουμε έναν έλεγχο αν έχετε όλοι φέρει τις ε, κάρτες σας και αν εκπροσωπούνται με τον σωστό αριθμό βουλευτών οι πολιτικές ομάδες. Γι' αυτό άρχεται ε, μια ψηφοφορία ελέγχου, δοκιμαστική. Λοιπόν, ε, οι σοσιαλιστές έχουν ένα περισσότερο, οπότε βγάζω εγώ τη δική μου κάρτα. Ωραία. 32 λοιπόν με δικαίωμα ψήφου είναι παρόντες, οπότε είναι όλα εντάξει. Περνάμε λοιπόν στο 15 ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Γένφελντ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με πολύ ευρία πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. 16. Και εδώ μία και μόνη ψηφοφορία. Είναι το θέμα της Κροατίας και της Κολομβίας και του Περού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εδώ εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία και εδώ συγχαίρουμε τον κύριο Φίσα. Τον κύριο Φίσας. 17. Αξιολόγηση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης, γνωμοδότηση. Λοιπόν, εδώ έχουμε πρώτα απ' όλα την συμβαστική 1. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 14 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 23, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25, υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εδώ να κάνουμε έλεγχο. Ψηφίζουμε την 25 άρχεται. Κατα... ε, πέρας, συγγνώμη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27, την οποία θα ψηφίσουμε σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 27 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και το τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται επίσης. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ψηφίζουμε επί της 29 άρχεται πέρας απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1. Υπάρχουν αντιρρήσεις ε, όσον αφορά την ψήφισή της. Ωραία. Άρα να ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Άρχεται πέρας εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική, άρχεται πέρας με 31 ψήφους υπέρ εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. ...18. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα ενός ιδιαίτερα μακροσκελούς και κουραστικού ε, τριλόγου... ...με πολλά δύσκολα σημεία και λάθη, αλλά εντάξει καταλήξαμε. Οπότε μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, άρχεται... 33 ψήφοι υπέρ εγκρίνεται ευχαριστώ πολύ οπότε έκλεισαν οι ψηφοφορίες μας σας ευχαριστώ πολύ περνάμε στο σημείο 19 για, τις, ε, για τη συμφωνία για τα προϊόντα τεχνολογίας της πληροφόρησης στα πλαίσια του ΠΟΕ. Το συζητήσαμε σύντομα και με την Επίτροπο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε όλοι να είστε συνεχώς παρόντες, αλλά εάν φεύγετε παρακαλώ να βγείτε ησύχω. Οπότε, τι έλεγα. Οπότε, συμφωνία ΙΤΑ, ITA. Και για το θέμα αυτό έχουμε έναν προσκεκλημένο μία προσκεκλημένη, την κυρία Άνκα Λίζα Σίλτ, που είναι σύμβουλος για θέματα εμπορικής και οικονομικής πολιτικής της εταιρείας Siemens. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Σίλντ. Πού είστε? Α, εκεί παρακαλώ. Ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους. Αν Σίλτε λέγομαι και δουλεύω στη Siemens εδώ για τις ε, κυβερνητικέ υποθέσεις ε, μου ζήτησαν ε, να μιλήσω λίγο για αυτή τη συμφωνία για τα προϊόντα τεχνολογίας. Ήμουν στην Γενέβη μέχρι χτες και ασχολούμαι με την συμφωνία, ασχολούμαι μέχρι τώρα με τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά άγαθα. Ξέρετε ότι έχουμε 350.000 υπαλλήλους παγκοσμίω, εκ των οποίων 200.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προϊόντα μας έχουμε το γεννήτριες, αυτόματες, αυτόματοι μηχανισμοί στη βιομηχανία, μεγάλες ιατρικές, ιατροτεχνικές συσκευές. Έχουμε ένα πολύ ευρύ φάσμα προϊόντων. Ό,τι έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση επίσης, 18.000 ε, Παραγωγού λογισμικών, προγραμματιστές λογισμικών έχουμε, οπότε ε, αυτή είναι μια βασική γραμμή δραστηριότητα για τη Siemens σε όλους τους τομείς. Για τις γεννήτριε, παραδείγματο χάρη, έχουμε αισθητήρε ε, που μα επιτρέπουν να παρακολουθούμε τη λειτουργία της, ε, ώστε με το πιο αποτελεσματικό τρόπο να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και να τοποθετήσουμε τι γεννήτριε μέσα σε ένα εργοστάσιο. Ε, είναι κύρια σημασία ε, τα εμπορικά ζητήματα για τη δραστηριότητά μας και θα σας δώσω τρεις λόγους ε, για τους οποίους θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή αυτή η συμφωνία για τα τεχνολογικά προϊόντα. Πρώτον, χορηγείται νέα πρόσβαση στην αγορά και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συμφωνία ATA. Πρόκειται για ένα πολυμερές πλαίσιο, δηλαδή ε, αυτό το συρφετό των διμερών συμφωνιών τελικά τον αφήνουμε πίσω μας, γιατί ξέρετε οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Είναι τόσες πολλές οι διμερείς ε, ε, συμφωνίες ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών που δημιουργεί πρόβλημα για μας. Λοιπόν, χορηγείται πρόσβαση στην αγορά, αυτό είναι πολύ θετικό για μας, μειώνονται οι δασμοί για, την, για τα ιατροτεχνικά προϊόντα στην Κίνα. Αυτό θα μας βοηθήσει πολύ. Απελευθέρωση σε ε, πολυμερές σχήμα πέρα από την ε, ενισχυμένη πρόσβαση στην αγορά με συστηματικό τρόπο ο πλευρά μάλλον συστήματο μπορούμε, όπω παρατηρήσαμε και στον Ναϊρόμπι, πήγα και εγώ ίδια εξάλλου εκεί, ε, όπου συζητήθηκε η σύναψη τη συμφωνία, μπορούμε λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε πλέον ότι τέτοιου αποτελέσματα χρειάζεται ο ΠΟΕ για να είναι θετική η ατμόσφαιρα και για να δείξουμε ότι ο ΠΟΕ μπορεί να έχει κεντρικό ρόλο. Όχι μόνο για τη διευθέτηση των διαφορών, κάτι που κάνει πολύ καλά, αλλά και για τον προσδιορισμό των κανόνων και απελευθέρωση του εμπορίου. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η συμφωνία. Ο τρίτος και τελευταίος λόγος που ε, στοιχειοδητεί τη σημασία της συμφωνίας αυτής είναι η δυνατότητα ε, να καθιστά δυνατή την ψηφιοποίηση. Όπως σας είπα για πολλές επιχειρήσεις και για τη δικιά μας κυρίως, είναι ε, καταλητικός αυτός ο παράγοντας για την ανταγωνιστικότητά μας. Τι επιτρέπουμε να κάνουν ε, στους πελάτες μας, παραδείγματος χάρη, να κάνουν ε, σε, ένα, σε μια κατασκευαστική μονάδα ένα, να κάνουν ένα ψηφιακό δίδυμο αυτής της εγκατάστασης. Δηλαδή, τι γίνεται αν δεν δοθεί αυτή η δυνατότητα. Πρέπει να σταματήσει η παραγωγή για να μπορέσει να δείτε αν θα, αν θα λειτουργήσει μια νέα μονάδα. Δηλαδή, κάνουμε ένα ψηφιακό, ένα εικονικό νέο έργο εργοστάσιο, ούτω ώστε σε επίπεδο μοντέλου να προγραμματίσετε τι αλλαγέ και προτού τι κάνετε να ξέρετε τι θα συμβεί. Ε, έτσι λοιπόν, σε πολλά προϊόντα που είναι απαραίτητα για την ψηφιοποίηση, για τους αισθητήρε παραδείγματο χάρη, αλλιώ παγώνουν συναλλαγές και ανέφερα τις αερογεννήτριες, ε, το χρησιμοποιούμε την ψηφιοποίηση σε πάρα πολλά προϊόντα, ούτως ώστε για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των προϊόντων να έχουμε περισσότερες πληροφορίες που στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πελάτες μας. Με τη συμφωνία λοιπόν έχουμε πλευρά συστήματος ε, τόνωση του ρόλου του ΠΟΕ, μας επιτρέπει την ε, ψηφιοποίηση, ε, και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Πρόεδρε, γιατί ήσασταν και εσείς στο Νεϊρόμπι με ένα κλιμάκι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δυστυχώς ε, δεν είχαμε πολλούς βουλευτές από άλλες περιοχές του κόσμου, όμως ε, έδωσε το παράδειγμα ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την ευρωπαϊκή διάσταση των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του ΠΟΕ. Θα σταματήσω εδώ και καλή επιτυχία για τη συνέχεια των συζητήσεων. Ευχαριστούμε. Ξέρουμε ποιο είναι το πλαίσιο τη συμφωνία ETA. Γνωρίζουμε τα ωφέλη της. Η εκπρόσωπος της Siemens θα επανέλαβε. Ξεκάθαρα υπάρχει ανάγκη και βούληση να προχωρήσουμε. Υπάρχουν βέβαια και χρονικοί περιορισμοί. Θα πρέπει η διαδικασία επικύρωση να έχει περατωθεί μέχρι πρώτη εβδόμου. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε άλλα προβλήματα. Είναι διαχειρίσιμε οι δυσκολίες πάντως. Τώρα μιλάω εγώ διότι δυστυχώ η συγκίτρια μας η κυρία Κίστ Χοντρόβολ δεν μπορεί να έρθει σήμερα. Συνέβη κάτι τραγικό στην οικογένειά της και ο Ντανή Κασπάρη θα την αντικαταστήσει. Α, και πριν, μέχρι πριν από 5 λεπτά ήταν εδώ. Να τον πάλι. Μπορώ να σταματήσω λοιπόν αυτή τη σύντομη ομιλία μου και να του δώσω το λόγο. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας ε, μιλήσω εκ μέρους της συναδέλφου που δεν θα μπορέσει να παραστεί σήμερα και θα σας διαβάσω τις σημειώσεις της. Λέει λοιπόν ότι η συμφωνία της επέκτασης της υφιστάμενης ε, συμφωνίας για τα τεχνολογικά προϊόντα πληροφορικής ε, είναι πολύ σημαντική. Ήταν η πρώτη συμφωνία που είχε ε, συναυθεί από τη σύσταση του ΠΟΕ και δεύτερον η συμφωνία αναμένεται να μειώσει το κόστος για τις καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και να υπάρχει ευρύτερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πληροφορικής. να σας δώσω και λίγο το ιστορικό. Αυτό εγκρίθηκε στη Σιγκαπούρη το 1990 1996, τέθηκε σε ισχύ ένα χρόνο αργότερα. Σήμερα υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντε που έχουν άρει δασμού σε τεχνολογικά προϊόντα όπως ψηφιακές κάμερες, τηλέφωνα κλπ. Αλλά έκτοτε ο τομέας τη πληροφορική έχει επεκταθεί και έπρεπε η συμφωνία να επεκταθεί σε νέα προϊόντα. Η απόφαση να επεκτείνουμε τα προϊόντα ξεκίνησε ε, το 2012 και τώρα έχουμε 54 μέλη του ΠΟΕ που διαπραγματεύτηκαν την διεύρυνση της συμφωνίας. Ε, κατάληξαν σε συμφωνία τον Ιούλιο πέρσι και την ενέκριναν οι Υπουργοί των Συμμετεχόντων Χωρών ε, φέτος ε, στην Υπουργική Διάσκεψη του Ναϊρόμπι υπομορφή δήλωσης για την επέκταση της ITA. Τι περιλαμβάνει η συμφωνία. Υπάρχουν συμβιβασμοί 201 ε, προϊόντων πληροφορικής, ημιαγωγού, συστήματα GPS, ιατροτεχνολογικά προϊόντα με μαγνητικές δυνατότητες και άλλα. Υπολογίζεται ότι έχουμε κύκλο εργασιών 1-3 ευρώ το χρόνο, επομένως πολύ μεγάλο τμήμα του παγκοσμίου εμπορίου φέτος. Ε, υπάρχουν δεσμεύσεις για όλα τα προϊόντα τα οποία έχουν κύκλο ζωής μέχρι και 7 χρόνια ε, έχουν προβλεφθεί περισσότερα, μεγαλύτερα διαστήματα για κάποια προϊόντα τα οποία μπορεί να χρειαστούν ίσως και ε, μεγαλύτερο χρόνο να προσαρμοστούν. Υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία καλύπτονται από την επέκταση και μετά από τις μειώσεις του διασμούς αναμένεται να ευξηθούν τα έσοδα. Συνολικά, η επέκταση της συμφωνίας έχει δυνατότητες να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και καινοτομία και επομένως ενθαρρύνει η συγγήτρια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, εγκρίνει αυτή τη συμφωνία και επίσης να σας πω ότι το, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορεύεται και με χώρες που δεν συμμετέχουν στη συμφωνία και θα υπάρχει δυνατότητα να υποφοληθούν ε, για τους δασμούς, αλλά δεν χρειάζεται να προσφέρουν τα ίδια ωφέλη για τα εισαγόμενα προϊόντα. Επομένως, για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απολαμβάνει πλήρως ε, των ωφελών, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα μέλη που θα ενταχθούν, ε, του ΠΟΕ, συγγνώμη, που θα ενταχθούν στη συμφωνία. Ωραία, να δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδης εισηγητές, η κυρία Μόσκα. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να υπογραμμίσω πόσο σημαντική ήταν η σύναψη αυτή τη συμφωνία, ε, η οποία είναι απαραίτητη λόγω τη ταχεία ε, τεχνολογική εξέλιξη 19 χρόνια μετά την πρώτη συμφωνία. Ευπρόσδεκτη συμφωνία και κρίμα που τη συζητούμε τόσο λίγο, διότι πρόκειται για μια συμφωνία η οποία μπορεί να προσφέρει πολύ μεγάλα ωφέλη και στους καταναλωτές και στους παραγωγούς και στην ευρωπαϊκή οικονομία εν γέννη και στους εταίρους μας. Κάποιες παρατηρήσεις μόνο. Και εγώ λοιπόν ελπίζω ότι θα ε, γίνουν σεβαστές όλες οι προθεσμίες ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν η συμφωνία. Ελάχιστες παρατηρήσεις. Καταρχάς και εγώ σημειώνω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει συμφωνία εντό του πολυμερού συστήματος, άρα ενισχύεται το σύστημα το οποίο εξακολουθούμε να προτιμούμε εμείς και ελπίζουμε και ότι και χώρες που σήμερα δεν έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία θα μπορέσουν να προσχωρήσουν στο μέλλον και να είναι και αυτές εταίροι. Επομένως να διευρύνουμε τα πιθανά ωφέλη. Δεύτερη παρατήρηση. Ελπίζουμε να μην χρειαστούν τόσο πολλά χρόνια για περαιτέρω επικαιροποίηση της συμφωνίας. Είναι θετικό λοιπόν το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί ήδη μια επικαιροποίηση το 2018 ίσως για να φτάσουμε και σε ένα μηχανισμό μόνιμης επικαιροποίησης ε, λόγω του συγκεκριμένου θέματος το οποίο άπτεται η συμφωνία που ξέρουμε ότι εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορεί να περιμένει οι εμπορικές συμφωνίες ε, να έχουν τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ της μίας επικαιροποίησης και της άλλης. Μια τελευταία παρατήρηση. Πολύ καλή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπεριλάβει και στις συζητήσεις ε, τη μείωση των μη δασμολογικών φραγμών στον τομέα αυτό και ελπίζουμε ότι το 2018 όταν θα ξαναξεκινήσει η συζήτηση ε, και η διαπραγμάτευση για το θέμα αυτό να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και κάποια θετικά αποφασιστικά βήματα και στον τομέα των μη δασμολογικών φραγμών. Ευχαριστώ πολύ. Για τους φιλελευθέρους, ε, η Μαρίτια. Ευχαριστώ. Είναι χρήσιμη αυτή η επικαιροποίηση της συμφωνίας γιατί μπορούμε πολλά να επιτύχουμε σε πολυμερές επίπεδο. Πρέπει να είμαστε απόλυτα ενήμεροι ότι έχει αλλάξει ο κόσμος. Πώς πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε ένα ανταγωνιστικό αποτέλεσμα αλλά πρέπει να επιδιώξουμε να επιβάλλουμε και τις αξίες μας. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε ένα σύστημα που να βασίζεται σε κανόνες Ελπίζω να πάμε γρήγορα. Ξέρουμε ότι μαζί με το θέμα του εμπορίου σε προϊόντα πληροφορικής η ανάπτυξη του ψηφιακού εμπορίου και των ψηφιακών υπηρεσιών σημαίνει γενικότερα ότι η οικονομία βασίζεται όλο και περισσότερο στι υπηρεσίε. Άρα σε όλε τι συμφωνίε που διαπραγματευόμεθα, τίζα, τίτυπη, οτιδήποτε άλλο, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε τις θεμελιώδεις αξίες ε, που είναι κοινέ σε όλους μας στην Ευρώπη και να ε, διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται χωρίς να παρεμποδίσουμε την ελεύθερη ροή πληροφοριών. Να ενθαρρύνουμε λοιπόν τις χώρες να ζητήσουν να μην ζητήσουν μάλλον ε, τα στοιχεία να συλλέγονται με τέτοιο τρόπο σε τοπικό επίπεδο που να δημιουργούν πρόβλημα για τον τρόπο λειτουργίες και καθορισμού των κανόνων και προδιαγραφών. Συμφωνώ με τη συνάδελφο Μόσκα ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το ρόλο που παίζει η τεχνολογία στο εμπόριο και ελπίζω να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση ως Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο και εμείς να παίξουμε ως Επιτροπή το ρόλο μας. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος, ο κύριος Μπούχνα. Συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν. Κάτι το οποίο πρόσεξα διαβάζοντας αυτή τη συμφωνία είναι ότι με αυτήν την ε, επέκταση της συμφωνίας χάνουμε την ε, βασική κατεύθυνση. Πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνουμε τώρα. Δηλαδή τα ψυγεία είναι και αυτά τώρα προϊόντα πληροφορικής ενώ άλλα δεν τα συμπεριλαμβάνουμε. Πρέπει να είμαστε πιο συστηματικοί σε τέτοιες συμφωνίες. Πρέπει να εξετάσουμε τι συμφωνίες δεν έχουμε ακόμη, ακόμη και τι θέλουμε να επιτύχουμε. Δεύτερον, κάτι που δεν ισχύει για αυτή τη νέα εκδοχή, αλλά γενικότερα. Παρατηρούμε ενίσχυση των μονοπωλιακών τάσεων στην αγορά σε αυτό το τομέα, από διάφορες απόψεις. Για ορισμένα προϊόντα παγκοσμίως υπάρχουν ένας ή δύο παραγωγοί. Αυτά τα θέματα πρέπει, ανεξάρτητα από αυτή τη συμφωνία, να τα εξετάσουμε. Αλλά θα επηρεάσει τέτοιου τύπου συμφωνίε οπωσδήποτε αυτή μα η εξέταση. Οπότε τίθεται το ερώτημα. Πώ θα αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη τάση δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Χαρμπάτη. Η ομάδα μας είναι εντελώ θετική. Χαιρετίζουμε την επικαιροποίηση σε αυτή τη συμφωνία για τα προϊόντα τεχνολογίας ε, πληροφορικής. Νομίζω ότι αυτή η επέκταση έχει μεγάλη σημασία γιατί το εμπόριο σε αυτά τα προϊόντα είναι ήδη 10% του παγκοσμίου εμπορίου και αυξάνεται. Χαιρετίζουμε ότι η συμφωνία αυτή η ITA ελέγχεται τακτικά για να είναι πάντα επίκαιρη θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε, να αυξήσουμε δηλαδή τον αριθμό των κρατών που συμμετέχουν και ελπίζω η Κομισιόν να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να ενθαρρύνουμε κάποια κράτη-μέλη να συμμετάσχουν, κάποια άλλα κράτη να συμμετάσχουν. Ε, πρόσεξα μια συγκεκριμένη διατύπωση της κυρίας Ρόρβολτ Λέει ότι σε ορισμένους τομείς αυξάνει ο ανταγωνισμός, αυξάνεται ο ανταγωνισμό. Αλλά ο κύριος Μπούχνερ αναφέρθηκε περισσότερο στον κίνδυνο μονοπωλίων. Ο ανταγωνισμός ε, σε μια ελεύθερη κοινωνία είναι θεμελιώδε συστατικό στοιχείο. Δεν είναι ανεπιθύμητη παρενέργεια, είναι κάτι το απόλυτα αναγκαίο γιατί ο ανταγωνισμός διασφαλίζει ότι δεν ανεβαίνουν πολύ τιμές και αν σκεφτώ τις συζητήσει που κάναμε χθε και σήμερα για το TTIP και για το CETA με εκπλήσει λιγάκι το πόσο αμυντικές είναι ορισμένες διατυπώσεις ορισμένων συναδέλφων. Ο κόσμος είναι ανοιχτό, άρα αυτό σημαίνει κινδύνους. Και αν κανείς δεν είναι διατεθειμένος να διατρέξει κινδύνους, αποκλείεται. Νομίζω ότι αν τα άτομα αυτά ήταν παρόντα και μπορούσαν να επηρεάσουν τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήταν κατά. Δεν υπάρχει κόσμος χωρίς κινδύνους και όποιος προσπαθεί να αποφύγει τους κινδύνους καταλήγει σε μια κλειστή και ε, βαλτωμένη κοινωνία. Αυτά ήθελα να τονίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Λουπέν. Ναι, αλλά κάποιε χώρε που δεν πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ λιγότερο στάσιμε από πολλέ χώρε τη Ένωση. Ε, εγώ θεωρώ το ότι είναι απόλυτα από άλλο κόσμο ότι έρχονται δύο εκπρόσωποι των μεγάλων ε, επιχειρήσεων να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους εδώ μέσα και να προτείνουν συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Αυτές οι συμφωνίες επιτρέπουν ε, να αυξηθούν οι ελεύθερες ε, συναλλαγές, ε, κάτι που το γουστάρεται ιδιαίτερα, χωρίς να ενημερώνετε τους λαούς. Δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνουν αυτές οι συμφωνίες. Είναι λιγότερο ορατές από τις συμφωνίες TTIP και με την Κίνα, αλλά παρόλα αυτά οι συμφωνίες αυτές έχουν ιδιαίτερα επιβλαβείς επιπτώσεις να κάνω μία παρομοίωση με μία άλλη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενα διαπραγμάτευση μεταξύ των 28 κρατών τη Ένωση και άλλων 16 χωρών. Κυρίε και κύριοι, σκέφτομαι ιδιαίτερα του πράσινου συναδέλφου. Θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θεωρείτε. Πολλέ χώρε θα είναι σε πολύ μειονεκτική θέση. Αν είναι υποχρεωμένε να χρησιμοποιούν αυτά τα οικολογικά προϊόντα για τι προμήθειέ του, αυτό σημαίνει ότι θα κατακλειστούν από ξένα τέτοια περιβαλλοντικά προϊόντα χωρίς δασμούς. Τι θα επιτύχετε? Θα καταστρέψετε τη δική μας ε, βιομηχανία αυτό το κλάδο προωθώντας τη χρήση περιβαλλοντικών προϊόντων. Αυτό έγινε και με τις ανανεώσιμες στη Γαλλία και σε ένα μεγάλο τμήμα της Ένωσης. Οι διάφοροι Κινέζοι παραγωγοί ε, εποφελήθηκαν από την αφέλειά σας και κατέκλυσαν τις αγορές μας. Ενώ στη δική τους εσωτερική αγορά προστατεύονται. Για άλλη μια φορά φοβάμαι ότι θα είναι άσχημο το ξύπνημα. Ευτυχώς οι λαοί αρχίζουν να ξυπνούν. Διαπιστώνουν με τρόμο τον ευρωπαϊκό εφιάλτη που ε, συνειδητά και ευσυνείδητα τους έχετε σερβίρει. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να αποφύγουν αυτόν τον ευρωπαϊκό εφιάλτη με κάθε νέο δημοψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ, και ο κύριος Μπορέλη τώρα τελευταίος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε γενικέ γραμμές δεν νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερε ενστάσεις για ένα τέτοιο θέμα. Έχω όμω κάποια ερωτηματικά για κάποιες κατηγορίες αγαθών που περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών των 200 προϊόντων που θα έχουν χαμηλότερους δασμού αγαθά τα οποία πιθανόν μπορεί να έχουν διπλή χρήση. Δορυφόροι, τμήμα δορυφόρων για τηλεπικοινωνίες, ε, ε, πηξίδες, ε, ε, και προϊόντα τα οποία μπορεί να επηρεάζουν την υγεία μας. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα για συγκεκριμένες ιατρικές, χειρουργικές, εκτινιατρικές εφαρμογές. Η άποψή μου είναι ότι η γενικότερη μείωση των δασμών, ναι μεν είναι θετική, αλλά δεν θα πρέπει να μειώνει και τις προδιαγραφές ε, στους τομείς αυτούς που ανέφερα παραπάνω και ούτε να ε, οδηγεί και σε απώλεια ε, και ζημίες για τους καταναλωτές. Ελπίζω λοιπόν για τα θέματα αυτά να μην μειώσει τα πάτη της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και τώρα Κομισιόν. Κορνέλη Σκίτσα. ο οποίο ήταν επικεφαλή των διαπραγματεύσεων από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη συμφωνία ITA. Ευχαριστώ. Είχα προετοιμάσει κάποιες σημειώσεις για να σας παρουσιάσω τα ωφέλη της επέκτασης συμφωνίας. Νομίζω όμως ότι τα είπατε εσείς πολύ καλύτερα από μένα οπότε μπορώ να είμαι σύντομος. Να αναφερθώ μόνο σε κάποια ζητήματα που ενδεχομένω παρλήθησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα ωφέλη. Οι εξαγωγές που καλύπτονται ε, επεσκελίζουν τις εισαγωγές δεν είναι ε, από μερκαντιλιστικής πλευράς ε, το σημαντικότερο, αλλά είναι μια παρηγοριά. Ε, πιο σημαντικό είναι το εξής. Έχουμε διάφορα επιθετικά ε, ε, προϊόντα κλειδιά σε βασικούς κλάδους Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία. Ε, Παραδείγματο χάρη τσίπ με πολλαπλές, πολλαπλών μερών, επίσης μηχανήματα που βασίζονται σε ημιαγωγούς, ε, ιατροτεχνολογικά προϊόντα που βασίζονται στις τεχνολογίες πληροφορίες, βιντεοπαιχνίδια. Σε όλους αυτούς τους τομείς είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί εμείς ε, και υπάρχει υψηλότατο αναπτυξιακό δυναμικό. Οπότε με τις νέες αγορές θα αυξηθούν την περαιτέρω εξαγωγές μας. Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα σημεία των καταλόγων είναι συστατικά μέρη που χρησιμοποιούνται για την ε, παρασκευή άλλων προϊόντων. Οπότε, ε, καταργώντας τους δασμούς για τις εισαγωγές αυτών των συστατικών, θα γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στη μεταποιητική μας βιομηχανία πέρα από τις εξαγωγές. Ε, και αυτό είναι σημαντικό όταν διαβάζετε την αποτίμηση της αξίας συμφωνίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δείτε πως ε, υπάρχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις και θα μας οδηγήσουν ε, σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα για την βιομηχανία μας και σε περισσότερες εξαγωγές και άρα και αυξημένο αριθμό θέσεων ε, απασχόλησης. Εξαιρούνται κάποια ευαίσθητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα και ε, μακροπρόθεσμα συμπεριλαμβάνονται άλλα, ούτως ώστε να έχει το χρόνο η βιομηχανία να προσαρμοστεί στην κατάργηση των δασμών. Ε, και φυσικά βασικό κομμάτι είναι οι δασμοί και τα μεγαλύτερα κέρδη που θα έχουμε προέρχονται από την Κίνα, διότι θα καταργήσει πολύ περισσότερους δασμούς η Κίνα για τις εισαγωγές από Ευρωπαϊκή Ένωση από το αντίθετο. Οπότε εμείς κερδίζουμε. Επίσης σημαντικό είναι ότι με τις χώρες με τις οποίες ήδη έχουμε τέτοια ΣΕΣ δεν θα υπάρχουν πιστοποιητικά και κανόνες προέλευσης. Ε, ε, σημαντική λοιπόν εξοικονόμηση από αυτή την πλευρά. να σχολιάσω και ένα-δύο σημαντικά ζητήματα που ανέφεραν και ε, οι βουλευτές, τα NTPs, Τώρα που ολοκληρώνονται οι, ολοκληρώνεται το τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων, έχουμε ακόμη μεγαλύτερο συμφέρον για τα NTBs και με τη βοήθεια της βιομηχανίας έχουμε καταλήξει μια νέα διαδικασία. Μόλις ήρθαμε από τη Γενέβη, γιατί κάναμε σύσκεψη ακριβώ για αυτό το ζήτημα, για τους μη δασμολογικούς, ε, μη εμπορικούς φραγμούς. Και Έχουμε και καλά νέα. Ε, κάποιες μικρότερες χώρες αποφάσισαν ε, να προσχωρήσουν συμφωνία. Μολδαβία, ε, Γεωργία, Μακάολα και κάποιες μεγαλύτερες ε, επί της αρχής συμφώνησαν ε, να προσχωρήσουν. Το Μεξικό, παραδείγματο χάρη, που ήταν και η μεγαλύτερη χώρα που απήχε από την IGA και η Χιλή. Ε, αυτά είναι πολύ καλά νέα και από 28 συμβαλόμενα μέρη της αρχικής ETA έχουμε περάσει τα 82, οπότε είναι πολύ καλές ε, οι ενδείξεις για την επέκταση της συμφωνίας και τον αριθμό των συμβαλωμένων μέρων. Ε, έχουμε καθυστερήσει, αλλά τηρούμε τις προθεσμίες. Στις 11 Απριλίου ενέκρινε το Συμβούλιο του Πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καταθέσουμε και στη συνέχεια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σχέδιο. Αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, τότε θα εγκριθεί απόφαση του Συμβουλίου και μετά από αυτό θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε εμείς κανονισμό για, τις, ε, για τους ε, Η προθεσμία στον τομέα του εμπορίου Προβλέπετε με κανονικά ε, κάπως μεγαλύτερη προθεσμία, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε μέχρι 1η Ιουλίου, εάν συνεργαστείτε κι εσείς. Εάν δηλαδή συνεργαστούν και τα τρία θεσμικά όργανα, είναι διαχειρίσιμη προθεσμία. Σας είμαστε ευγνώμενος για την υποστήριξή σας, για την υλοποίηση αυτών των στόχων που έχουμε θέσει. Ευχαριστούμε. Πρόεδρος. Δεν απαντήσατε όμως στις, απαν... στις ερωτήσεις του κυρίου Μπορέλη για τα προϊόντα διπλής χρήσης, παραδείγματος χάρη. Θέλετε να το σχολιάσετε. Πολλά προϊόντα έχουν δει χρήση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς. Υπάρχουν όμως ξεκάθαροι κανόνες και αρμόδιες επιτροπές. Δεν νομίζω ότι η κατάργηση του δοσμολογικού τέλους θα επηρεάσει την κατάσταση για αυτά τα αγαθά. Ε, πιο πολύ είναι θέμα εισαγωγικών αδειών και αποτροπή εξαγωγών, ώστε να μην καταλήξουν τα προϊόντα σε λάθος χώρες. Ε, το ύψος των δασμών δεν επηρεάζει ε, σημαντικά την κατάσταση, Πρόεδρος, και εγώ το ίδιο πιστεύω, όμως πρέπει να συμπεριλάβουμε τον τομέα της πληροφορικής ε, στον κανονισμό περί προϊόντων διετής χρήσης. Νομίζω είναι βασικό στοιχείο και το έχουμε συζητήσει. Είχαμε, περιμέναμε μία πρόταση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί αυτού μετά το καλοκαίρι. Ωραία. Η συγκήτρια λείπει, οπότε δεν έχει άλλα ε, σχόλια. Η καταληκτική προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι 25 Απριλίου. Στην Επιτροπή θα ψηφίσουμε στις 24 Μαΐου και μπορούμε στην πρώτη ολομέλεια του Ιουνίου να ε, ψηφίσουμε για την έκθεση που δίνει την συγκατάθεση του Κοινοβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούμε και με το χρονοδιάγραμμα που εσείς μας επιβάλλετε, δηλαδή να έχουμε ολοκληρώσει τα πάντα μέχρι 1η Ιουλίου. Ευχαριστώ. Τώρα ε, πάμε πίσω στο σημείο 11. Θυμάστε ότι αναβάλαμε την εξέταση του ζητήματος αυτού είναι η αναθεώρηση των τεχνικών κανόνων ε, από τον οργανισμό της ε, Γενέβης ίσως να μην είναι τόσο σεξι αυτό το θέμα αλλά είναι αυτό το οποίο θέλουμε να ε, επιτύχουμε για τη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών αφορά τα οχήματα, ε, τα τροχοφόρα οχήματα και την αναθεώρηση των οχημάτων και των τμήματων που μπορούν να εφαρμοστούν σε ε, οχήματα. Θέλουμε λοιπόν να ξαναβάλουμε στην, στο κέντρο της προσοχής μας τα θέματα αυτά και σε τι βαθμό αυτά τα θέματα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σε διμερείς εμπορικές συμφωνίες. Η ομάδα 29 στη Γενέβη είναι η αρμόδια για την ενημέρωση τέτοιων συμφωνιών. Υπάρχει το 58 αυτή η συμφωνία, έχουν γίνει δύο αναθεωρήσεις. Τώρα είναι η τρίτη αναθεώρηση για να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία αυτό που επιδιώκουμε είναι να υπάρχει ένας τύπος έγκρισης ε, για τα ε, οχήματα και να υπάρχει περισσότερη συνέπεια στην ε, λήψη αποφάσεων. Έχει αυξηθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία από τα 2 τρίτα στα 4 πέμπτα. ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη περισσότερη άποψη των μειοψηφιών από αυτήν την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών. Εθνών. Είναι λοιπόν χρήσιμη αυτή η προσπάθεια, αυτός ο τρόπος λειτουργίας και για να έχουμε υψηλό επίπεδο προδιαγραφών και για να αποφεύγουμε άσκοπες επικαλύψεις ε, προσπαθειών και κόστους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τη συζήτηση με τις ΗΠΑ ε, για τα αυτοκίνητα, αν και οι δύο συμμετείχαμε ε, ενεργώς ε, στις συζητήσεις της Τεχνικής Επιτροπής της, Γενέ... της Οικονομικής συγγνώμη, Επιτροπής της Γενέβης για τα θέματα αυτά. Θα μπορούσαμε να επιλύσουμε έτσι πολλά προβλήματα. Κάλεσα την Κομισιόν να μας εξηγήσει τη σχέση μεταξύ αυτής της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων και της διμερής εμπορικές συμφωνίες. Και από ό,τι βλέπω εδώ είναι παρόν ο αναπληρωτής τμήματάρχης για να μας παρουσιάσει τα θέματα αυτά. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι υπάλληλο. Ε, ο αναπληρώτρια τριματάρχης δεν θα μπορέσει να παραστεί. Σας ευχαριστώ λοιπόν για το σχέδιο σύστασης και σας ευχαριστούμε γι' αυτό και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε τις απόψεις μας για την ε, διεθνή ρυθμιστική συνεργασία. Είναι πολύ σημαντική αυτή, ε, εν γέννη, αλλά κυρίω για το τομέα τη αυτοκινητοβιομηχανίας. Βοηθά την δημιουργία θέσεων εργασία και ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα και την περιβαλλοντική προστασία. Θα ήθελα να σα παρουσιάσω το βασικό πλαίσιο επί τη οποία ε, επί του οποίου συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιτύχει αυτή τη ρυθμιστική συνεργασία με τρίτες χώρες και την εναρμόνιση των ε, κανονισμών για τα οχήματα ως πρότυπο για τους διεθνείς κανονισμούς για τα ε, ταξινόμηση των οχημάτων. Επίσης θα σας πω και λίγα λόγια για τη Συμφωνία του 1958, το οποίο είναι θέμα του σχεδίου απόφασης. Γιατί είναι κρίσιμη σημασία λοιπόν η διεθνή ε, συνεργασία, κυρίω στον τομέα τη αυτοκινητοβιομηχανία, στα θέματα αυτά. Υπάρχουν διαφορέ ε, στι ρυθμιστικέ απαιτήσει, ε, διπλασιασμό απαιτήσεων και αλληλοεπικάλυψη, που ορισμένε φορέ δημιουργούν μη δεσμολογικού φραγμού στο εμπόριο. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσει δίνουν κονδύλια σε αναποτελεσματικέ μεθόδου προσαρμογή ή ταξινόμηση, που δεν έχουν κανένα περιβαλλοντικό όφελο και προστατεύουν απλώ τι σε εγχώριες αγορές. Ίσως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια για επενδύσεις ε, και έρευνα για να δημιουργήσουμε ε, νέες θέσει εργασίες. Επίσης υπάρχει ε, όφελος ε, δημιουργεί οικονομίας κλίμακας και άρει του φραγμούς στο εμπόριο. Γι' αυτό και ακριβώ η διεθνή ρυθμιστική συνεργασία είναι τόσο σημαντική και ιδίω στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Όπως αναφέρεται επίσης στο σχέδιο σύστασης, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ένας από τους κινητήριους μοχλούς της ευρωπαϊκής οικονομίας και σε θέματα ΑΕΠ και σε θέματα θέσεων εργασία και οικονομικά. Είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε έρευνα και ανάπτυξη. Επίσης, η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ταυτόχρονα και παγκόσμια βιομηχανία. Ε, έχει σχέση με παγκόσμιες αλυσίδες αγοράς και αυξάνεται η επιρροή της ε, σταδιακά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όρημη αγορά, αλλά υπάρχουν κάποιες χώρες και περιοχές οι οποίες γίνονται όλο και πιο σημαντικέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 80% της ανάπτυξης στον τομέα θα γίνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στις αναδυόμενες οικονομίες. Ο ευρωπαϊκός τομέας αυτοκινητοβιομηχανίας έχει μεγάλη επιρροή στο διεθνές εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθαρός εξαγωγέας ε, αυτοκινήτων και ανταλλακτικών και ε, γενικότερα είναι θετικές οι τάσεις. Υπάρχει μας στα οχήματα το 2014 που ήταν 95 ε, εκατομμύρια ευρώ, δις ευρώ, συγγνώμη, η παρούσα κατάσταση όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Η διεθνής ε, ε, ανταγωνιστική κατάσταση εντείνει τις ε, τάσεις και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της ρύθμισης. Πρέπει να εμπερδίσουμε στις παραγωγές αυτοκινήτων και να μειώσουμε τις εντάσεις από τον ανταγωνισμό, κυρίως μέσω της άρσης μη φραγμών. Όπως σας είπαμε, πιστεύουμε ότι η παγκόσμια ρυθμιστική συνεργασία είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους μη δεσμολογικούς ε, φραγμούς. Επίσης, βοηθά την οδική ασφάλεια και το περιβάλλον και έχουμε περισσότερο φιλόδοξες ε, ρυθμιστικές πρακτικές ε, και προδιαγραφές σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως για τις χώρες οι οποίες υστερούν ένα καλό παράδειγμα για να δείξουμε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία αυτή για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας είναι η έγκριση σε επίπεδο UNICE ενός νέου μοντέλου για τις εκπομπές αυτοκινήτων, ε, τα νέα τεστ WLTP για τα ελαφρά οχήματα. Αυτό έγινε χάρη σε συνεισφορά εμπειρογνωμόνων και δεδομένων που συλλέχθηκαν παγκοσμίω. Αυτή η νέα διαδικασία είναι πιο αντιπροσωπευτική της ε, πραγματικής ε, ε, δυνατότητας εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και έτσι μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές και να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Επομένως, για τη συνεργασία αυτή θα σταθώ στο συμφωνία της Γιούνισε. Όπως σας είπα προηγουμένως, ένα κατάλληλο πλαίσιο είναι το πλαίσιο που έχουμε από τα Ηνωμένα Έθνη του 1950 8 ε, λέγεται WP29. Εκεί είναι συμβαλόμενο μέρος η Ευρωπαϊκή Ένωση και ηγείται ε, των εργασιών για δύο συμφωνίες. Η πρώτη είναι η συμφωνία του 59 για την ανάπτυξη οχημάτων και όταν ε, το προβλέπουν τα συμβολέμωνα μέρη υπάρχει και αμοιβαία αναγνώριση αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει 129 κανονισμούς από τους 136 και η βασική μας εταίροι είναι η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Νότια Κορέα και η Αυστραλία. Το Μάιο του 2016 η Ιαπωνία θα εφαρμόζει 66 κανονισμούς. Η δεύτερη συμφωνία, η Συμφωνία του 98, είναι πιο παγκόσμια συμφωνία, περιλαμβάνει τι ΗΠΑ, την Ινδία και την Κίνα για την ανάπτυξη των λεγόμενων τεχνικών παγκόσμιων κανονισμών. Μέχρι τώρα υπάρχουν 16 εγκεκριμένοι τεχνικοί κανονισμοί που δεν προβλέπουν και αμοιβαία αναγνώριση. Οι αποφάσει λαμβάνονται μέσω συνένεση και όχι με πλειοψηφία 2 τρίτων. Ε, για την συμφωνία του 59 και τη μεταρρύθμισή σας, ε, ε, τη μεταρρύθμισή σας θα σας πω αργότερα, αλλά νομίζω ότι γίνονται προσπάθειες για βελτίωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία και όπως πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος, είναι πολύ σημαντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένα έγγραφο τριμερές για, με συστάσεις για το πώς θα μπορέσει να γίνει πιο καλή αυτή η συνεργασία που θα εγκριθεί τον Ιούνιο. Προωθούμε επίσης ε, το ρυθμιστικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και στις διμερείς μας ε, επαφές που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως κύριε Πρόεδρε. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο διαρθρωμένου βιομηχανικού ή ρυθμιστικού διαλόγου, για παράδειγμα με την Κίνα, με την Ιαπωνία ή με τη Ρωσία. Και στο πλαίσιο των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. Σε αυτές τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που συνάφτησαν πρόσφατα υπάρχει και ένα συγκεκριμένο παράρτημα στον τομέα αυτό για να υπάρχει σύγκληση ε, προς ε, τους κανονισμούς ε, του UNICE. Και επίσης υπάρχουν και ενεξελέξει διαπραγματεύσεις, όπως για παράδειγμα με την TTIP, ε, ε, με την Ιαπωνία και τις χώρες της ΑΣΕΑΝ, στις οποίες θέλουμε να το συμπεριλάβουμε. Έρχομαι στο τελευταίο τμήμα τη παρέμβασή μου, την αναθεώρηση για αυτή τη ρυθμιστική συνεργασία της Συμφωνία του 1958. Όπως σα είπα, Βάσει του φόρουμ του UNEC, η συμφωνία του 1958 είναι συμφωνία κομβική για την εναρμόνιση. Πρόκειται για πολύ σημαντικό εργαλείο και τα συμβαλόμενα μέρη αυτόματα ε, σημαίνει ότι δέχονται στην αγορά τους αυτοκίνητα, οχήματα, ανταλλακτικά ε, και εξαρτήματα τα οποία συμμορφούνται προς τον κανονισμό. στα πλαίσια των εργασιών για την πλήρη έγκριση τύπου οχημάτων μπορεί να υπάρχει και διεθνή ε, εναρμόνιση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πάει πέρα-πέρα. Στον ε, ε, κανονισμό για την ασφάλεια που εγκρίθηκε το 2009 εφαρμόζονται κάποιες οδηγίες του UNICE απευθείας ως ευρωπαϊκό δίκαιο. Και δεν περιορίζεται μάλιστα αυτή η συμφωνία στα συμβαλόμενα μέρη. Οι κανονισμοί αυτοί ισχύουν και σε χώρες που δεν έχουν προσυπογράψει, όπως την Κίνα και την Ινδία το γεγονός ότι παρέχεται και από χώρε που δεν έχουν συμφωνήσει για τη συμφωνία σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση των αυτοκινήτων σε αυτές τις αγορές. Παρά το γεγονό ότι η Συμφωνία του 1958 αποδείχθηκε ότι είναι πολύ καλό εργαλείο για τη ρυθμιστική συνεργασία, κατέστη σαφέ τα τελευταία χρόνια ότι πρέπει να τη μεταρρυθμίσουμε. Και η μεταρρύθμιση ε, έγινε για δύο κυρίω λόγου. Πρώτον, για να αυξήσουμε την ελκυστικότητα τη Συμφωνία του 1958, κυρίω με χώρε που έχουν αναδεόμενε αυτοκινητοβιομηχανίε, και εδώ έχουμε την αλλαγή που ανέφερε ο Πρόεδρο. Και το δεύτερο είναι να έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα είναι κατάλληλος και εύρωστος για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στο μέλλον σε μια συνεχώς εναλλασσόμενη αγορά στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, διαθέσει πόρους για τη μεταρρύθμιση αυτή και είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Βασιζόμαστε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει θετική άποψη για την αναθεώρηση του WP29 τον Ιούνιο και να συνεχίσει η Συμφωνία του 58 να αποτελεί πρότυπο για τη ρυθμιστική συνεργασία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Ε, geschätzte ähm, Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που είναι απόλυτα σαφές από αυτή την παρουσίαση είναι ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση τα πάμε πολύ καλά στην ρυθμιστική συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια. Χαιρετίζω αυτό στο οποίο καταλήξαμε, είναι περαιτέρω βελτίωση. Γιατί έχουμε αυτές τις προδιαγραφές. Θα ήθελα να τονίσω ότι τις έχουμε για να συμμετάσχουν όσο δυνατόν περισσότεροι. Αυτό ισχύει και για το TTIP και για πολλές άλλες συμφωνίες. Όπως εάν χώρες όπως η Ιαπωνία ή η Νότια Κορέα θέλουν να έχουν ισότιμες σχέσεις μαζί μας, καλό θα ήταν να συμμετέχουν σε αυτές τις συμφωνίες. Δεν χρειάζεται λοιπόν ε, να έχουμε τόσο πολλές διαφορετικές προδιαγραφές. Και στο παρελθόν ως Επιτροπή έχουμε επανειλημμένα πει ότι μας στέλνουν προτάσεις αυτοί οι οργανισμοί, είδαμε τι περιέχουν, είδαμε αν συμβαδίζουν με το ρυθμιστικό πλαίσιο που έχουμε ως Ένωση και κατόπιν ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο έχουμε βεβαιώσει ε, ότι θέλουμε αυτές τις συμφωνίες, αλλά βέβαια αν θεωρούσαμε ότι δεν συμβαδίζουν θα το απορρίπταμε. Αυτό αποδεικνύει πώς μπορεί να λειτουργήσει η ρυθμιστική συνεργασία, δηλαδή κάθονται μαζί οι ειδικοί, εξετάζουν ε, τις προτάσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη και την εθνική νομοθεσία που υπάρχει ήδη στα διάφορα κράτη του κόσμου και παρόλα αυτά οι προτάσεις που κάνουν είναι αποδεκτές από τους περισσότερους. Αλλά κάνουν προτάσεις. Δεν αποφασίζουν. Εμείς αποφασίζουμε ως Κοινοβούλιο μαζί με τον συνομοθέτη, το Συμβούλιο. Αυτό θέλω να πω. Για την ομάδα μας θα στηρίξουμε και αυτή την πρόταση όπως την προτείνει ο εισηγητής και παραλαμβάνω ότι είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα που πρέπει να αξιοποιήσουμε και ανοιχτά να πούμε στους πολίτες μας ότι η ρυθμιστική συνεργασία δεν είναι κακή, δεν είναι επικίνδυνη, αλλά αντίθετα μας επιτρέπει στον ανταγωνισμό με τις άλλες χώρες του κόσμου και είναι καλό το ότι υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος, δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ε, βεβαίως να αναφερθώ και σε αυτά που είπε ο κύριος Κασπάρη και στο ψήφισμά μας για το TTIP Αναφέραμε το αποτέλεσμα του UNEC και της Ομάδας Εργασίας 29 που είπαμε ότι είναι ένα λειτουργικό μοντέλο δημοκρατικού ελέγχου της ρυθμιστικής συνεργασίας. Το είπαμε εκπεφρασμένα. Νομίζω ότι είναι ένα σαφές μήνυμα ότι μπορούμε και με τους ε, έξω κοινοτικούς εταίρους μας να έχουμε άλλες μεθόδους ρυθμιστικής συνεργασίας και αυτό το παράδειγμα είναι καλό. Και δεν αποδεχόμεθα ενδεχομένω κάποιε άλλε μορφέ ρυθμιστική συνεργασία. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 22 Δευτέρα, τρέχοντος. Και το Μάιο νομίζω θα ψηφίσουμε. Το Μάιο, μάλιστα. Ωραία. Οπότε να περάσουμε στο σημείο 20. Και αυτό είναι συναρπαστικό. Είναι παρουσίαση Είναι η παρουσίαση λοιπόν μιας ε, έκθεσης που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως για την επίπτωση των, οικονομικ... των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στις ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου της Ένωσης και σχετίζεται με τη συζήτηση για τις διαρροές από το Παναμά, τα Panama Leaks. Είναι λοιπόν πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Το Πανεπιστήμιο του Χρόνιγχεν, το οποίο εκπονεί αυτή τη μελέτη, έχουμε, έχουμε εδώ ορισμένου ερευνητές και ερευνήτριες. Θα τους δώσω το λόγο. Αλλά θέλω να καταστήσω σαφές ότι είναι ακόμη σχέδιο μελέτης, δεν είναι ακόμη το τελικό κείμενο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, αξιότιμοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη που εκπονήσαμε, όπως σωστά είπατε, στο Πανεπιστήμιο του Χρόνγκεν μαζί με το Ινστιτούτο ΑΣΕΡ ε, των ε, Κάτω Χωρών Έχουμε ένα τετραμέρες κλιμάκι εδώ, Όλκα Κιτσένκο, δίπλα μου, από το Χρόνιγεν, από το Άσερ, ο Ντάβου Γιάνσιτς και από το Χρόνιγεν και πάλι η Άντζη και υποφαινόμενος από το Άσερ. Σωστά είπατε, Πρόεδρε, αυτή η έκθεση ε, θα, πρέπει να χτενιστεί ακόμη. Ε, είναι εξαιρετικά επίκαιρη όμως για θέματα φοροαποφυγής και διαφυγής. Ε, είναι μεγάλο το δημόσιο ενδιαφέρον για τα εμπορικά ζητήματα επίσης, όχι μόνο για την TTIP ε, και επειδή είμαι ο Ολλανδός δεν μπορώ παρά να αναφερθώ και στην Συμφωνία Σύνδεση με την Ουκρανία. Στον ΟΣΑ και στην Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης συζητούνται αυτά ακριβώς τα ζητήματα την FATF. Έχω και διαφάνειες. Δεν μπορώ όμως να προχωρήσω. Μπορείτε να βάλετε το επόμενο, την επόμενη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Σας μίλησα λίγο για τα συμφραζόμενα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να διευρύνει ε, τις, ε, τους στόχους της για τις εξωτερικές σχέσεις και το εμπόριο με τρίτες χώρες με προώθηση του κράτους δικαίου βιώσιμης ανάπτυξης και πολύ φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη συνθήκη της Λισαβόνας έχει ήδη οριστεί αυτό και στην στρατηγική εμπόριο για όλους του 2015. Είναι επίκαιρο το ζήτημα επίσης διότι πρόσφατα ανέλευε πρωτοβουλία σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομοθεσία για ζητήματα φοροαποφυγής, διαφυγής, διαφάνειας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ταυτόχρονα με την απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών ορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε εμπορικές συμφωνίες και τη νέα νομοθεσία για την νομιμοποίηση εισόδου και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, αναλύσαμε το περιεχόμενο 5 FTAs, 5 σες τέτοιων συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών και τις διατάξεις για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για τη φοροαποφυγή, διαφυγή και νομοποίηση εσόδων ε, και την, αναλύσαμε την εφαρμογή των συμφωνιών στις τρίτες χώρες. Αυτό ήταν το νομικό ε, κομμάτι της μελέτης ε, και μετά παρουσιάζουμε και μία ανάλυση των επιπτώσεων, πρακτικών επιπτώσεων στο εμπειρικό κομμάτι της μελέτης και στο τέλος συνάγουμε και συμπεράζουμε και συστάσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Όπως σας είπα, το νομικό, στο νομικό κομμάτι έχουμε τις ε, εκθέσεις ε, ε, ανά χώρα, έξι χώρες, γιατί μία ευθεία καλύπτει και την Κολομβία και το Περού, δύο χώρες δηλαδή. Βλέπετε στη διαφάνεια τι βρήκαμε. Κατά μέσο όρο δεν είναι αρκετά ισχυρή η διατύπωση γιατί μιλάμε για best endeavors, καλύτερη ε, προσπάθεια για την ανάληψη δράσεως κατά της νομοποίησης εσόδων παράνομες δραστηριότητες ε, και αυτή η διατύπωση δεν αποτελεί επαρκές κίνητρο για τους εμπορικούς μας για να αναλάβουν την απαιτούμενη δράση. Επίσης, ε, πολλές ε, χώρες ε, έχουν ένα καλό, επιχάρτουν νομικό πλαίσιο, αυτό δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα, είναι τυπικά εντάξει. Τα βασικά αποπορίσματα όμως στο νομικό κομμάτι κάλυψαν μάλλον ε, μας οδηγούν στα συμπεράσματα ότι δεν ε, λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι, ε, αυτές οι διατάξεις στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και Επίσης δεν συμμετέχει επαρκώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαδικασίες. Εμείς πιστεύουμε σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνεται στις εκθέσεις για την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών και στο μέτρο που υπάρχουν πληροφορίες για όλες αυτές τις ε, χώρες, ακόμη και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των συμφωνιών ε, για το ασθενές ε, κράτος δικαίου, για την εφαρμογή που χωλαίνει, υπάρχουν, υπάρχει ενημέρωση από επίσημες πηγές και θα σας δώσουμε και παραδείγματα. Πέρα στην επόμενη διαφάνεια. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Όλγα, τη συνάδελφό μου. Θα ήθελα να, να σας παρουσιάσω τα συμπεράσματα του εμπειρικού τμήματος της αξιολόγησης των συμφωνιών υπό το φως της νομοθεσίας για τη φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και νομοποίηση εσόδων παράνομους δραστηριότητες. Τι εννοηθήκαμε λοιπόν σε αυτή τη μελέτη. Εάν η απελευθέρωση του εμπορίου ανάμεσα στην Ένωση και τις τρίτες χώρες κυρίως για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εντείνει το, τον κίνδυνο ε, νομοποίησης αυτών των παράνομων δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν ούτως ή άλλως αυτές οι χώρες. Τα, ποια είναι τα ευρήματα της έκθεσης που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Γενικά γίνεται αποδεκτό ότι οι παράνομες χρηματοπιστωτικές από τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, είναι πολύ σημαντικές και αυξάνονται διαρκώς παρότι δεν έχουμε επακριβή στατιστική αποτίμηση αυτών των παρανόμων χρηματοπιστωτικών ροών. Γνωρίζουμε ε, ότι είναι πολύ μεγάλο το εύρος του φαινομένου και Μπορείτε να περάσετε στην μεθεπόμενη διαφάνεια, γιατί έχουμε κάποια δεδομένα στατιστικά. Άλλη μία. Ωραία, ευχαριστώ. Όπως δείχνουν τα δεδομένα, ε, και ε, ε, ε, η βασικός οργανισμός για την εκπόνηση στατιστικών στοιχείων για τις παράνομες χρηματοπιστωτικές αέρες και την ανάλυση τους δείχνει πως το Μεξικό και η Νότια Αφρική είναι οι δύο πρώτες στον κατάλογο στη σειρά ως προς τις παράνομες χρηματοπιστωτικές ροές στον κόσμο των αναπτυσσομένων χωρών. Βλέπετε μετά ακολουθούν η Κίνα, Ρωσία. Και τα την τελευταία ετία βλέπουμε ένα βασικό μια ε, κεντρική τάση αύξησης ε, των παρανόμων σωματοπιστωτικών ροών, διαρκούς αύξησης αυτών των ροών. Ε, υπάρχουν λοιπόν και άλλες αφρικανικές χώρες που ακολουθούν ε, από τη θέση 7 και μετά. Και βασιζόμενοι σε αυτά τα δεδομένα βλέπουμε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες στην περίπτωση ε, μας ε, Κολομβία, Περού, πέρα από το Μεξικό δηλαδή και την Νότια Αφρική και τη Σερβία που είναι, έχει μεταβατικό καθεστώς, ε, υπάρχει σοβαρή απειλή για επανομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το θέμα είναι πώς ακριβώς αυτή η απειλή συνδέεται με τις ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά πόσο εντείνεται η απειλή. Λόγω αυτών των συμφωνιών μπορείτε παρακαλώ να επανέλθετε στην πέμπτη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Εκεί που λέει ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων. Εδώ. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ε, στατιστικά και το στατιστικά δεδομένα που να αποδεικνύουν πέραν κάθε αμφιβολία σε σχέση αιτιατού ε, ε, ανάμεσα στις ε, ε, Συμφωνίες Ελευθερών και την αύξηση των παρανόμων χρηματοπιστωτικών ροών. Όμω είναι ισχυρή η τάση και το στοιχειοθετείται αυτό από τα δεδομένα που συλλέξαμε ότι οι συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι προαναφερθήσει χώρε ουσιαστικά ε, εντείνουν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τους άλλους αυτές τις χώρες για την νομιμοποίηση εσόδων παρανόμων δραστηριότητων. Τρεις συμπαράγοντε πρέπει να συνεκτιμήσουμε. υπό το φως αυτών των ευρημάτων. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις σε σχέση με το σημαντικό βαθμό ανοίγματο μετά την υπογραφή τέτοιων ΣΕΣ, τέτοιων συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών και ακόμη σημαντικότερα οι παράνομες χρηματοπιστωτικές ροές από τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ήδη σημαντικές και διαρκώς αυξανόμενες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο ε, και μπορεί ε, να δειχθεί σε βασικό συμπέρασμα, δηλαδή είμαστε ελκυστικό ο για τη νομοποίηση των παρνόμων δραστηριοτήτων ροών προερχομένων από αναπτυσσόμενε ε, χώρες. το ίδιο το άνοιγμα τη αγορά εντείνει ε, τον κίνδυνο αναρωτιόμαστε εμείς, ε, θεωρούμε ότι ισχύει, ε, ευσταθεί αυτό, εντείνεται ο κίνδυνος ε, κυρίως διότι ε, υπάρχει μια ουσιαστική ισχυρή απειλή που αντιμετωπίζουν αυτές οι χώρες στον τομέα του, της νομιμοποίησης εσόδων και είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί οι θεσμοί, ε, οι φορείς μάλλον που μπορεί να χρησιμοποιηθούν γι' αυτό λόγο στις δυτικές χώρες. Δεν δίνω παράδειγμα. Ε, για το Μεξικό. Οι χρηματοπιστωτικοί τέτοιοι φορείς σε αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως ε, μάλλον στις δικές μας χώρες, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ε, για τους καταθέτες ε, από το Μεξικό την τελευταία δεκαετία. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα και αφορά μόνο το Μεξικό. Εξίσου σημαντικό είναι να τονίσουμε και αυτό ε, μας έκανε εντύπωση κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της ε, μελέτης. Οι ροές αυτές ε, οι χρηματοπιστωτικές δεν χρησιμοποιούν μόνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δηλαδή δεν ξεπλένεται αυτό το χρήμα χρησιμοποιώντας μόνο το ε, χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ε, με την ε, ε, εσφαλμένη τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών βασιζόμενο στο εμπόριο γίνεται πλέον ως επιτοπλίστων τη σήμερα ημέρα η νομιμοποίηση εσόδων παρανόμων δραστηριοτήτων. Βλέπουμε πώς μπαίνουν εμφανώς οι ροές μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και ξαναβγαίνουν ε, επί τη βάση εμπορικών συναλλαγών από την πίσω πόρτα τα ίδια χρήματα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι παράνομες χρηματοπιστωτικές ροές που λαμβάνουν αυτή τη μορφή εισρωών και εκροών έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση ε, στην οικονομία των αναπτυσσομένων χωρών, κυρίως ως προς το αναπτυξιακό του δυναμικό και είναι παράδοξο το ότι ε, υπάρχει μία συμφωνία και βλέπουμε τα ποσά των παρανόμων χρηματοπιστωτικών ροών που έρχονται από τι αναπτυσσόμενες χώρες πολλές φορές υπερβαίνουν το ύψος της αναπτυξιακής βοήθειας ε, που λαμβάνουν από τον ανεπτυγμένο κόσμο αυτές οι χώρες ε, και βάση ε, του οργανισμού για την, το Παγκοσμίου Οργανισμού για την Χρηματοπιστωτική Ακαιρεότητα με στοιχεία 2013 για κάθε δολάριο αναπτυξιακή αναπτυξιακής βοήθεια που παίρνουν αυτές οι χώρες έχαναν 10 δολάρια αυτές ε, οι χώρες ε, σε παράνομες χρηματοπιστωτικές δροές. 1 προς 10. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω Χρειαζόμαστε και άλλες στατιστικές κυρίως ή να επικεντρωθούμε στα αίτια των ε, παρανόμων οικονομικών ροών που επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και η μελέτη μας δείχνει ότι το γράμμα του νόμου είναι εντελώ άλλο από το πώς εφαρμόζεται ο νόμος, γιατί η αδυναμία στην εφαρμογή του νόμου είναι πολύ σημαντικές για τις, για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως μια επιφύλαξη. Μπορεί να θεωρείτε ότι εμείς νομίζουμε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι η ρίζα του προβλήματος για την καταπολέμηση της νομοποίησης προϊόντος ε, εγκλήματος. Βεβαίως παίζουν μεγάλο ρόλο οι αδυναμίες των αναπτυσσόμενων χωρών αλλά και οι έλεγχοι στις δυτικές χώρες, ιδιαίτερα στην Ένωση δεν είναι επαρκής και επιδεινώνουν την κατάσταση. Ένα παράδειγμα. Η τράπεζα HSBC που έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει εμπλακεί επανειλημμένα <clears throat> σε σκάνδαλα για τέτοια νομιμοποίηση εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ε, νομιμοποίησης ε, προσόδων εγκληματικών καρτέλ ναρκωτικών, ένα με βάση το Μεξικό και ένα με βάση την Κολομβία. Τώρα για τις ε, συστάσεις. Για να δούμε μερικά αριθμητικά στοιχεία. Πόσες καταδίκες έχουμε για τέτοια παράνομη νομοποίηση. Νομοποίηση μάλλον προσόδων ε, εγκλήματος. Βλέπετε εδώ τα στοιχεία. Παράδειγμα, Περού. Μηδέν καταδίκες. Για καμία δραστηριότητα τέτοιου τύπου. Ούτε τότε ούτε παλιότερα, γιατί το μηδέν είναι από παλιά. Είναι μηδέν και μηδέν και μηδέν. Συγγνώμη, ε, αφορούσε την Κορέα εκ το Περού. Αφορούσαν την Κορέα τα στοιχεία αυτά. Μια αναπτυγμένη χώρα όπως η Κορέα λοιπόν δεν καταφέρνει να έχει ε, καταδίκες. Πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτές τις χώρες λοιπόν. Να περάσουμε στο τελευταίο, τελευταία διαφάνεια. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε για να εφαρμοστούν αυτοί οι στόχοι για κράτος δικαίου, βιώσιμη ανάπτυξη κτλ. πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη πιο σοβαρά στις εμπορικές σχέσεις. Πρέπει να επιχειρήσουμε να ασκήσουμε πίεση, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε συμπερίληψη τέτοιων θεμάτων στις εμπορικές συμφωνίες, στα συστήματα των μελετών αντικτύπου να περιλαμβάνονται τέτοια κριτήρια το συζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά υπάρχουν ακόμη πολύ σοβαρέ αδυναμίε. Γιατί οι μελέτε αντικτύπου δεν είναι έτοιμε όταν καταλήγουν οι διαπραγματεύσει. Και το TTIP είναι ένα καλό παράδειγμα, κραυγαλαίο παράδειγμα. Δεν είναι ακόμη έτοιμη αυτή η μελέτη αντικτύπου. Αναμένεται το Σεπτέμβριο, που θα είναι πολύ αργά για να παίξει ρόλο στι ίδιε τι διαπραγματεύσει. Και για να μπορέσει να εκφραστεί επί των ε, πορισμάτων αυτή τη μελέτη και το Κοινοβούλιο. Βεβαίως χρειάζεται γενικά περισσότερη διεθνή συνεργασία. Θέλουμε μια πιο ευρεία προσέγγιση για την εμπορική πολιτική και να εφαρμοστεί αυτή η πιο ευρεία προσέγγιση ούτως για να συνδεθούν οι στόχοι στην εμπορική πολιτική με την, τους ευρύτερους στόχους της Ένωσης για καλή διακυβέρνηση. Επίσης ε, προτείνουμε επειδή θέλουμε να αυξηθεί και η δημοκρατική αποδοχή είναι ένας στόχος αυτός γιατί η κοινή γνώμη θέτει και πολλά μη εμπορικά θέματα στα πλαίσια αυτά πρέπει να παίξει αυξημένο ρόλο το Κοινοβούλιο στην επιτήρηση της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και σε σχέση με αυτά που είπε και η συνάδελφός μου πολέμηση της πολιτικής καθορισμού καταχρηστικών τιμών στο διεθνές εμπόριο. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την κατάρτιση και την τεχνική βοήθεια στις ε, χώρες ε, με τις οποίες έχουμε σχέση, ούτω ώστε να εφαρμόζεται καλύτερα ο νόμος. Και τέλος, αλλά επίσης πολύ σημαντικό, θέλουμε να συμμετάσχουν και οι αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου, τα γραφεία του Κοινοβουλίου στην επιτήρηση της ε, παρακολούθησης ε, της καταπολέμησης της νομιμοποίησης προϊόντος εγκλήματος. Και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο τα νομοθετικά κείμενα που έχουμε και η ίδια η συνθήκη αλλά και οι νόμοι των ε, εταίρων μας οι νόμοι αυτοί να εφαρμοστούν στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη αυτή. Τα στοιχεία που μας δώσατε, τα στατιστικά στοιχεία νομίζω είναι εύγλωτα και οι συστάσεις σας βεβαίως. Ορισμένες φορές ε, ίσως πρέπει κάποιες ε, συστάσεις να είναι λίγο πιο συγκεκριμένες. Θέλει κανείς το λόγο Ε, ε, εσείς, Γιούντι, ήσασταν πρώτοι, μετά ο κύριος Μπούχνερ και η Ήμα. Ευχαριστώ. Ως ε, εισηγήτρια για την οδηγία κατά της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων που είχε ε, πονήσει πριν από κάποια χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα παρακολούθησα όλα αυτά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα ήθελα να ξέρω αν απαντάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελέτη σήμερα ή θα απαντήσει κάποια στιγμή. γιατί θα ήθελα να θέσω και σε αυτούς ερωτήσεις. Ναι, βεβαίως έχει εκπρόσωπο της Κομισιόν εδώ και μπορεί να απαντήσει, αλλά συνήθως ε, κάνουμε τη συζήτηση μεταξύ μας και μετά απαντά. Τίποτα, απλώ αναρωτιέμαι αν μπορώ να θέσω ερωτήσεις και προς την Κομισιόν. Διότι, διαβάζοντας κανείς την έκθεση, διαπιστώνει για παράδειγμα ότι η περιφερειακή εφαρμογή των προτύπων των Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών ε, στην Κολομβία και στο Περό δεν έχουν επικαιροποιηθεί από το 2008. Σας το λέω αυτό ε, διότι αν το ξέρουμε και έχουν ε, με συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με αυτές τις χώρες, ξέρουμε ότι καθυστερούν κατά ένα-δύο χρόνια την εφαρμογή. Γι' αυτό και ακριβώς και έγινε πλήρης αναθεώρηση της οδηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση των παρανόμων εσόδων. Τι κάνουμε λοιπόν στη διαπραγμάτευση για τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου ώστε να φροντίσουμε οι εταίροι μας να υποχρεωθούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα δράσης ε, για τις υποχρεώσεις αυτές. Είμαστε και μέσω της συζήτησης για τα Panama Papers και αποφασίσαμε από πλευράς Κοινοβουλίου να κάνουμε έρευνα επί του θέματος. Πώς ε, βλέπουμε τις συμφωνίες Ελευθερού ε, Εμπορίου υπό αυτό το πνεύμα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν ε, οι συνάδελφοι, αλλά σήμερα είχε έρθει ο Καμπέκ εδώ, μιλούσε στην Επιτροπή Ανάπτυξης ως πρόεδρος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των παρανόμων ροών χρημάτων από την Νότια Αφρική, που το ανέφεραν και οι ερευνητές. Και δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι δεν είμαστε συνεπείς ε, προς τις πολιτικές μας ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ως προς τους ε, συντάκτες της μελέτης. Τις είδαμε τις συστάσεις σας, αλλά τι δυνατότητα βλέπετε εσείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουν ε, πιο ε, αυστηρή διατύπωση στις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου επί του θέματο αυτού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Κύριος Μπουχτερ. Ευχαριστώ πολύ. Μία σύντομη ερώτηση. Μας κάνουν συστάσεις σε εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο. Στις διαπραγματεύσεις ε, που κάνουμε με πολλές χώρες για συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου όπως το Μεξικό θα ληφθούν υπόψη αυτές οι συστάσεις στο Μεξικό και παρόμοια είναι η κατάσταση και σε άλλες χώρες. Είναι καλή η νομοθεσία που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα εάν τηρεί το, αλλά δεν τηρεί την νομοθεσία. Με τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου μπορούμε μέσω συμπερίληψης ε, τέτοιων ρητρών θα είχαμε μία δυνατότητα να αλλάξουμε μία κατάσταση που η αλλαγή της θα ήταν προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Άρα, καθήκον μας θα πρέπει να είναι τους προσεχείς μήνες στις διαπραγματεύσεις να συμπεριλάβουμε αυτές τις συστάσεις. Θα γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Άλλη μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Ναι, ναι, θα πάρει το λόγο η ΙΜΑ. Βεβαίω με τα θέματα πολέμης διαφθοράς ήδη ασχολούμε, θα έχουμε την στρατηγική για το εμπόριο όπου το αναφέρουμε και θα αποστείλουμε, τώρα εκπονούμε μία επιστολή προς την Κομισιόν όπου τονίζουμε ότι πρέπει ακριβώς τα θέματα <clears throat> διαφθοράς να αντιμετωπιστούν και να συμπεριληφθούν ε, για τη νέα μας στρατηγική για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις. Η Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι αντίστοιχη με του κύριου Μπούχνερ. Μάλλον απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή εξυγχρονίζουμε την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό που αναφέρει ως τρίτη χώρα και μάλιστα με αυξανόμενες τάσεις για παράνομες ροές χρημάτων και θα ήθελα να ξέρω σε ποιο βαθμό μπορούν να ληφθούν μέτρα προκειμένου να βοηθήσουμε να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ε, να συγχαρώ τους συντάκτες της μελέτης ε, για την παρουσίασή τους και θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε να μου πείτε γιατί με εντυπωσίασε η εξέλιξη της Ρωσίας στη στην νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, αυξάνει με αλματώδεις ρυθμούς η Κίνα. Ε, η Ρωσία έλαβε κάποια μέτρα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ε, δεν ε, αποτελούν πραγματικά απάντηση σε συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων. Uh, Και εγώ να ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, ο κύριος Σόλτς. Δύο ερωτήσεις προς τους συντάκτες. Μας παρουσιάζετε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες χώρες. Το πρόβλημα βέβαια αφορά πολύ περισσότερες χώρες. Και μετά τι. Αν για παράδειγμα βλέπουμε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, είναι προφανές ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα Μπορείτε να εμβαθύνετε στη μελέτη αυτού του τόσο περίπλοκου ε, θέματος και άλλο. και τι μπορούμε να περιμένουμε εν είδη συμπερασμάτων για την επόμενη χρονιά όταν θα συζητήσουμε τα θέματα εμπορίου και συμφωνίες ε, με τις χώρες αυτές. Και το αυτό ισχύει φυσικά και για άλλες αφρικανικές χώρες, κεντροασιατικές χώρες κλπ. Και, και φυσικά και εμάς. Και αυτή είναι η δεύτερη ερώτησή μου. Διότι έχουμε το ξέπλυμα, μεν, αλλά από την άλλη ε, τίθεται και θέμα φοροδιαφυγής σε κάποιο βαθμό. Η φοροδιαφυγή, αν ε, τη συγκρίνεται με τα διαβόητα Panama Papers, ο Παναμάς είναι στην τρίτη θέση. Στη δεύτερη ε, χώρα είναι ε, θέση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία στην 8η. τι σημαίνει αυτό για το πρόβλημα το οποίο περιγράφετε στη μελέτη σας και τι θα πρέπει εμείς να λάβουμε υπόψη ενό συνομοθέτε όταν αναφερόμαστε σε χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε ε, και σε θέματα τα οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε στι ε, εμπορικέ συμφωνίε ή στι επενδυτικέ συμφωνίε, ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο ή τουλάχιστον να το περιορίσουμε. Και κάτι ακόμα, ίσως δεν κατάλαβα καλά βέβαια, σε ένα από τα συμπεράσματα στις συστάσεις ε, για τους όρους αναφερθήκατε σε αυτό το, το, τους όρους που πρέπει να θέσουμε. Μπορείτε να πείτε λίγα παραπάνω από αυτού. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν τώρα. Πολύν, wine Selling, για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ και την υπηρεσία μελετών του Κοινοβουλίου που παρήγγειλε αυτή την μελέτη και θέλουμε να δούμε και την τελική της ε, εκδοχή γιατί ασχολείται με θέματα που είναι προτεραιότητες ε, του πολιτικού μας θεματολογίου και συζητούμε πολλά ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, που σχετίζονται με την νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος, την φοροδιαφυγή και φόρο αποφυγή. Φυσικά, η μελέτη προσπαθεί να δει τη σύνδεση μεταξύ της ε, ε, απελευθέρωσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και παρανόμων χρηματικών ροών. Και ναι, δεν υπάρχει σαφή στατιστική διασύνδεση, αλλά καταλήγει σε σημαντικές ε, διαπιστώσεις ε, για τα θέματα αυτά. Πολύ ενδιαφέρον. Και η σύσταση για την καταπολέμηση του καθορισμού υπερβολικά υψηλών τιμών στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια διτή προσέγγιση. Δηλαδή πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε και τη δική μας εσωτερική πολιτική για την εφαρμογή της, τέταρτη της τέταρτης οδηγίας για την νομιμοποίηση του εγκλήματος. Είναι κάτι που το κάνει αυτή τη στιγμή η Γενική Διεύθυνση για θέματα δικαιοσύνης. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και την νομιμοποίηση μέσω δραστηριοτήτων εμπορίου. Για τα θέματα αυτά η Κομισιόν ακόμη φέτος αλλά και του χρόνου θα καταλήξει σε ορισμένα πορίσματα για το πώς μπορούμε εντός της Ένωσης να το αντιμετωπίσουμε και επίσης πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών. Παράλληλα, οι συνάδελφοί μας που ασχολούνται με τα τελωνία το εξετάζουν. Αυτή τη στιγμή γίνονται πολλές μελέτες για να ενισχύσουμε την ε, καταπολέμηση του καθορισμού λοιπόν καταχρηστικών τιμών όσον αφορά την φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, νομιμοποίηση είπα ότι και αυτά είναι υψηλές προτεραιότητες και λόγω των προσφάτων διαρών εγγράφων από τον Παναμά το εξετάζουμε μαζί με τους συναδέλφους ε, με έναν ε, τρόπο ενιαίο ως υπηρεσίες για να σας πω τι γίνεται γενικότερα και πώς συνδέεται με αυτά που κάνουμε για τις συμφωνίες εμπορίου. Ε, θέλουμε λοιπόν να καταπολεμήσουμε την ε, φοροδιαφυγή στα πλαίσια και της εξωτερικής μας στρατηγικής. Θέλουμε λοιπόν η προσέγγιση μας να ε, καταλήξει στην κατάρτιση ενός ε, καταλόγου όπου οι φορολογικές αρχές ε, δεν συνεργάζονται και δεν εφαρμόζουν διεθνείς προδιαγραφές όπως για παράδειγμα ανταλλαγή στοιχείων. Στα πλαίσια αυτά είναι σαφές ότι θα μελετήσουμε τον τρόπο εφαρμογής των προδιαγραφών καλής διακυβέρνησης ούτως ώστε να δούμε πώς εφαρμόζονται ρήτρες που συμπεριλαμβάνονται σε διεθνεί συμφωνίε και συνεργαζόμαστε φυσικά με άλλε υπηρεσίε πολύ στενά. Επιπλέον, την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν ενέκρινε μια νέα πρόταση για την τρομοποίηση της οδηγίας για την ε, υποβολή εκθέσεων αναχώρα για τις ε, μεγάλες πολυεθνικές. Και ιδιαίτερα για χώρες ε, που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους καταλόγους που προανέφερα. Τρίτη επίσης σημαντική πλευρά, όπως ήδη αναφέρθηκε από ορισμένου από τους παρόντες ευρωβουλευτές, είναι η εφαρμογή της αναθεωρημένης ε, οδηγίας για την ε, νομιμοποίηση προϊόντος ε, εγκλήματος, ιδιαίτερα για το ποιος είναι ο ουσιαστικός ιδιοκτήτης που επωφελείται από, για παράδειγμα, ε, συγκεκριμένες ε, δραστηριότητες και επίσης για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ορισμένων χωρών που έχουν αδυναμίες ε, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης με βάση τις συστάσεις της συγκεκριμένη Task Force. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό. Γιατί αυτή η Task Force για την δράση στο χρηματοπιστωτικό τομέα είναι ο σημαντικότερος φορέας που ασχολείται με αυτά τα θέματα και η Κομισιόν για τα θέματα αυτά θα εγκρίνει μια περαιτέρω προσέγγιση της Ένωσης για αυτό. Επιπλέον, σε πολλά διεθνή φόρα όπως το G20 προωθούμε τα θέματα αυτά και μέσω των μηχανισμών που υπάρχουν λοιπόν όπως είπα αυτό το Financial Action Task Force Και επίσης ε, οι ερευνητές αναφέρθηκαν στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες τρίτων χωρών. Και για το θέμα αυτό πρέπει να πούμε ότι η Επιτροπή βοηθάει, δίνει τεχνική βοήθεια για να δημιουργηθούν οι δυνατότητες. Αναφέρθηκε ήδη αυτό. Όλα αυτά ήδη γίνονται. Βέβαια πρέπει να δούμε πώς μπορούν να βοηθήσουν και οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, πώς μπορούν να συμπληρώσουν αυτά που ήδη κάνουμε, όπως σωστά ήδη επισημάνθηκε. Η ανακοίνωση εμπόριο για όλους που ενεκρίθη τον περασμένο Οκτώβριο τονίζει ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες να αντιμετωπιστούν οι επιθετικές τακτικές μεταφοράς κερδών των πολυεθνικών και να προωθήσει διεθνείς προδιαγραφές για διαφάνεια και χρηστή διακυβέρνηση. Όπως ήδη εξάλλου υπόθηκε, οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου ήδη αναφέρονται στην χρηστή διακυβέρνηση και για θέματα φορολογικά και για θέματα νομιμοποίησης προϊόντος εγκλήματος και στα πλαίσια της εξωτερικής στρατηγικής ήδη αναφέρθηκα, είμαστε σε φάση απολογισμού για το πώς εφαρμόζονται αυτές οι αρχές χρηστής διακυβέρνησης που είναι ήδη στα κεφάλαια για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Γιατί πολλά έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουν βελτιωθεί οι διεθνείς προδιαγραφές μέσω του ΟΣΑ και του G20. Οπότε εξετάζουμε πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί συγκεκριμένα μέσω αυτών των ρητρών. Είναι μια δουλειά που ήδη γίνεται. Επίσης ε, συζητήσατε σήμερα το ότι οι προσεγγίσεις αυτές είναι οι προσεγγίσεις ε, της βέλτιστης δυνατής προσπάθειας. Best endeavor όπως λέγεται και αν θα έπρεπε να γίνουν περισσότερο προϋποθέσεις. Το σκεφτήκαμε πολύ. Όπως είπαμε υπάρχουν ήδη μηχανισμοί που, που λειτουργούν. για να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ανεπάρκειες. Και θα αντιμετωπιστεί περαιτέρω το θέμα αυτό και μέσω των καταλόγων αυτών που θα εγκρίνει η Ένωση. Όπου υπάρχουν λοιπόν ανεπάρκειες, θα υπάρξει μηχανισμός κάλυψης και ε, γίνονται συνεχώς και αναθεωρήσεις του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων. Άρα πρέπει να δούμε. Χρειάζεται ανάγκη να κάνουμε και άλλα μέσω των ε, εμπορικών συμφωνιών. Υπάρχουν αυτές οι ρήτρες χρηστής διακυβέρνησης που είναι μια καλή σύνδεση μεταξύ αυτών των προσπαθειών και αυτών που περιέχουν οι εμπορικές συμφωνίες. Και υπάρχουν διάφορα φόρα όπου ασχολούμεθα ήδη με, τον, με την νομιμοποίηση παρανόμων. Και επίσης βέβαια πάντα ε, είμαστε υπέρ ε, συνεργασίας για την αντιμετώπιση αυτών των ε, θεμάτων. Είπαμε για παράδειγμα ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη ρυθμιστική συνεργασία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στα πλαίσια των συμφωνιών εμπορίου ή αλλού για να ασκήσουμε πιέσεις ε, επί των εταίρων μας και να πιέσουμε για να εφαρμοστούν οι κανόνες για την νομιμοποίηση παρανόμων προσόδων. Και η μελέτη στα πλαίσια αυτά κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση για τις αναπτυσσόμενες και τις αναπτυγμένες χώρες. Και νομίζουμε ότι πρέπει να βρούμε μηχανισμούς συνεργασίας. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Γιατί οι αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις για να αποκτήσουν ε, το αναγκαίο προσωπικό, τις αναγκαίες ικανότητες για να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Και στα πλαίσια του δικού μας ε, καθεστώτος για το θέμα αυτό εντός της Ένωσης είναι καλό να έχουμε τέτοιους καταλόγους. Όπως προσπαθούμε να κάνουμε και για την φόρο διαφυγή και αποφυγή. Υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν διαδικασίες υποεκπώνηση για να βοηθήσουμε τις χώρες να δημιουργήσουν το δυναμικό για να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα. Και αν οι χώρες αυτές δεν συνεργαστούν και δεν εφαρμόσουν τις προδιαγραφές, τότε υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Για να συνοψίσω. Η στρατηγική μπορεί για όλους Βεβαίως, στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας, προβάλλει ότι οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου δεν πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα. Συνδέονται με την ε, χρηστή φορολογική διακυβέρνηση και την καταπολέμηση της ε, νομιμοποίησης. Πρέπει να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για αυτά. Επίσης αναφερθήκατε και στη σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Βεβαίως, το τονίζω και αυτό. Γιατί δεν το αναφέρει η μελέτη. Όπως ξέρετε, έχουμε δεσμευθεί στην ανακοίνωση αυτή να προτείνουμε φιλόδοξα μέτρα για τη μελλοντική καταπολέμηση της διαφθοράς και σχετίζεται βεβαίως με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης. Για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για το ποιο είναι ο ουσιαστικό κάτοχο. Είναι κάτι που το αναφέρει και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση διαφθορά. Στον τομέα αυτό θέλουμε να προωθήσουμε μέσω των συμφωνιών ελευθερών αυτές τις αρχές. Κάτι άλλο, τελικό, Αν εξετάσουμε όλες μας τις εμπορικές συμφωνίες με όλους τους εταίρους βλέπετε ότι δεν τις εξετάζουμε μονομένα θέλουμε να βοηθήσουν την αντιμετώπιση των παρανόμων οικονομικών ροών. Και άρα αναμένουμε και τη δική σας στήριξη στις συνομιλίες με τους εταίρους μας για να υπάρξει συνειδητοποίηση και να καταλάβουν ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουν για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα. Τέλος! Υπήρχαν και μερικά άλλα θέματα για συγκεκριμένες εμπορικές συμφωνίες για την Κολομβία και τις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις με το Μεξικό. Για την Κολομβία. Είναι ήδη λειτουργούσα συμφωνία. εάν υπάρχουν, εάν υπάρχουν ανεπάρκειες για τους κανόνες που περιέχει για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης, τότε πρέπει να το δούμε. Υπάρχουν κατάλογοι, είπα, που εκπονούμε. που ε, ε, πρέπει να εφαρμοστούν σε συνδυασμό με τις συστάσεις ε, της Task Force για τα θέματα αυτά. Εάν υπάρχουν ε, αδυναμίες στην περίπτωση της Κολομβίας, αυτοί είναι οι μηχανισμοί για να τους αντιμετωπίσουν. Για το Μεξικό. Είμαστε ακόμη σε προπαρασκευαστική φάση για την επικαιροποίηση της υπάρχουσας συμφωνίας αλλά προτείνουμε να συμπεριληφθούν ρήτρες σε αυτή τη νέα συμφωνία, την επικαιροποίηση δηλαδή, για καταπολέμηση της διαφθοράς. Και θα δούμε και τη σύνδεση με, τον, με την νομιμοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε για την εντελεχέστατη απάντηση. Θα δώσω το λόγο στους ερευνητές. Ευχαριστούμε για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να απαντήσουμε το μέγιστο αριθμό ερωτήσεων. Από τις πιο σημαντικές είναι κατά τη γνώμη μας τι πρέπει να γίνει για να υπάρχει μια ισχυρότερη διατύπωση μέσα στις ε, συμφωνίες Ελευθερών εμπορίου. Είναι δυνατό, η συνάδελφος θα το σχολιάσει λεπτομερέστερα, αλλά για να δούμε τι κάνουν οι Αμερικανοί ε, για αυτό το ζήτημα βλέπουμε ότι υπάρχουν σαφέστατες ρήτρες στις εμπορικές συμφωνίες με τις ίδιες χώρες σε πολλές περιπτώσεις. Τι λένε, έχουμε πέντε ελεγκτές τώρα και θα έχουμε 500 ε, σε λίγα χρόνια. Δηλαδή τόσο συγκεκριμένες είναι οι διατάξεις και τόσο συγκεκριμένοι πρέπει να είσαστε ε, ούτως ώστε να επιβάλλετε καλύτερα η νομοθεσία. Ακόμη και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι κάνει άλμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι συμπεριλαμβάνει κεφάλαια βιώσιμη ανάπτυξη σε καλύτερη παρακολούθηση, εποπτεία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτά τα παραδείγματα αυτά σε μια πρώτη φάση και ο Νταρφέρ θα μας συνεχίσει, θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Εφτά ε, σχόλια θα ήθελα να, να, αναφέρω, ε, ε, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σχολιάσω την, τη θεώρηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις πολιτικές ε, συνδυάζοντας την ε, με τη, τα σχόλιά μας ε, για τη, με την εμπορική πολιτική της 29 Ιανουαρίου 2016. Ζητά επανεκτίμηση ε, της εμπορικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα φορολογικά ζητήματα και η ίδια η Επιτροπή αναφέρει ότι είναι η πιο διατύπωση σε πολλές περιπτώσεις, ε, παραδείγματος χάρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα. Και άρα δεν είναι σαφώς επιτυχημένα τα αποτελέσματα, διότι αρνούνται αναλάβουν δέσμευση κάποιοι εταιρικοί. Η ίδια η Επιτροπή προτείνει ένα screening με ένα πίνακα βαθμολόγηση, μια εξέταση δηλαδή και σύγκριση, ούτω ώστε να υπάρχει αιρεσιμότητα με την ακόλουθη μορφή. Οι επενδύσει ε, στα ταμεία θα απαγορεύονται στο μέτρο που δεν πληρεί η χώρα τα διεθνή πρότυπα για την ε, καταπολέμηση τη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Αυτά για την Επιτροπή. Τώρα α περάσουμε στι δικέ μα συστάσει μια σταδιακή απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυτό είχαμε κατά νου. Τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα απελευθερώσει αν προϋποθέσεων τις χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίες. Θα είναι συνάρτηση της εφαρμογής των διεθνών προτύπων αυτή η απελευθέρωση. Δηλαδή η πιερωσιμότητα τρόπον την ε, τι πρέπει να κάνουμε με την Ανατολή, θα, τη Ρωσία θα την αφήσω στον συνάδελφο, αλλά θέλω να μιλήσω για την Κίνα που είναι ακόμη σημαντικότερη. Το 2013 οι ε, αρχές ε, για την ε, καταπολέμηση της φοροποφυγής, φοροδιαφύγης και νομοποίησης ε, ε, εκτίμησαν την αξία στα 150 δις, ε, ενώ για τη Ρωσία ήταν 120 δις. Ε, το Δεκέμβρη πέρσι είχαμε ένα ψήφισμα για τις σχέσεις με την Κίνα, όμως εκεί δεν αναφέρθηκε η φοροαποφύγη, φοροδιαφύγη και το ξέπλυμα χρήματος, ε, μιλούσαν μόνο για τις κρατικές ενισχύσεις. Λοιπόν, είναι σημαντικό και αυτό να είναι θέμα συζήτησης και να μην αποφεύγουμε το βασικό αυτό ζήτημα. Τρίτον, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ανατολή αλλά και στη Δύση. Η Επίτροπος για το Εμπόριο, η κυρία Μάλστρομ, ήταν νωρίτερα εδώ και η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν είχε διατάξεις για την απελευθέρωση των υπηρεσιών σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Όμως από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών και από τον ΩΣΑ έχω στοιχεία που δείχνουν πως 83, 83 από τις βασικές ε, εταιρείε έχουν θηγατρικές σε φορολογικές παραδείσους. Ένα τρεις στα Κέιμαν παραδείγματος, ένα τρεις δολάρια ε, σε στοιχεία ενεργητικού. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό και τα θέματα τα φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και τα λοιπά πρέπει να τα βλέπουμε και με ανε... ανεπτυγμένες χώρες. Όχι μόνο με αναπτυσσόμενε. Τα έγγραφα του Παναμά δείχνουν ότι δεν μιλάμε για οργανώσεις, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείε που διαπράττουν αυτές τις αξιόπινες πράξεις, αλλά και ε, μεμονωμένα άτομα. Θα πρέπει να το τονίσουμε ε, και αυτό και πάλι να το ξαναπώ αφορά και τις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τώρα, ε, έλλειψη συνοχής στις πολιτικές. Νότια Αφρική, ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα. Ε, τονίζουμε το θέμα της Νότιας Αφρικής, διότι ανήκει στην Παναφρικανική Ένωση, στην Αφρικανική Ένωση της Νοτιού και ε, εκεί απευθύνονται ε, κρίσει κατά της Νοτιού ε, διότι συνάπτει συμφωνίες γενικευμένων προτιμήσεων με άλλες τρίτες χώρες πλήττοντα έτσι τις υπόλοιπες αφρικανικές χώρες αυτή τη Ένωση. Έκτο σημείο. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ανατολικών χωρών ή των λιγότερων ανεπτυγμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τρόπο που ε, αντιμετωπίζουν αυτά τα δύο προβλήματα. Ένα πολύ επιτυχημένο ε, παράδειγμα είναι αυτό της ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σερβία 2,2 δις και χρηματοδότηση από πλευρά της Ένωσης 90% και σχεδόν 10% το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, συγχρηματοδότηση λοιπόν κράτησε χρόνια και ε, καταλήξαμε σε μια πρώτη έκθεση για την καταπολέμηση αυτών των δύο φαινομένων στη Σερβία όπου τονίζεται η σημασία του να δίνουμε στις χώρες σε καθεστώς μετάβασης ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες και γενικότερα σε εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωσης επί συνεργασία συγγνώμη, ακόμη και σε διοικητικό επίπεδο. Τέλος, να τονίσω κι εγώ Νομίζω πέρσι ήταν ένα λεπτό, ναι, ναι, τον Ιούνιο του 2015 δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα κατάλογο ε, ε, αρχών τρίτων χωρών που δεν συνεργάζονται για θέματα φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής. Ακόμη και εκεί δεν είναι πλήρης ο κατάλογος. Φερρυπίν, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία δεν αναγνωρίζουν αυτό τον κατάλογο. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε και μια συνοχή σε αυτά που κάνουμε και να ε, ε, είναι πλήρη η ενημέρωση. Θα δώσω τώρα στο Χάινιχ, το συνάδελφο εδώ. Ναι. Μια πολύ σύντομη απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή για τη Ρωσία και τις τάσεις στη Ρωσία που δημιουργεί λογικά ερωτηματικά λόγω και του πίνακα που είδατε σε κάποια από τις διαφάνειες. Στη σελίδα 15 του σχεδίου έκθεσής μας μπορείτε να δείτε ότι στον κατάλογο των ε, παράνομων ε, οικονομικών ροών από τις 10 ε, πρώτες χώρες η Ρωσία είναι στη δεύτερη θέση. Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μελετήσαμε μόνο πέντε χώρε όμω, μόνο πέντε συμφωνίε ελευθέρωσης λαγών. Επομένω, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα συμπεράσματά μα σε σχέση με τι άλλε χώρε. Πρέπει να τονίσω βέβαια ότι επιλέξαμε αυτές τις χώρες και αυτές τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών γιατί είναι χώρες οι οποίες έχουν διαφορετικά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και επίσης τις επιλέξαμε και ως χώρες οι οποίες διασφαλίζουν ένα ε, συγκεκριμένο βαθμό γεωγραφικής κάλυψης. Επομένω θέλουμε να έχουμε σημαντικά στοιχεία από χώρες. Δεν θα πω λεπτομέρειες για την κατάσταση στη Ρωσία, αλλά να σας πω ποιο είναι το γενικότερο συμπέρασμά μας. Υπάρχει αύξηση των παράνομων ε, ε, οικονομικών ροών, ε, υπάρχει σχέση με την απελευθέρωση η οποία εφαρμόζεται και υπάρχει διαφορετικός νόμος στο γράμμα του νόμου και διαφορετικά πράγματα εφαρμόζονται στην πράξη, που είναι και μία από τις συστάσεις μου. Τα συστήματα επιβολής του νόμου στις χώρες πρέπει να εφαρμόζονται και ε, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θέλαμε να ε, προτείνουμε τεχνική συνδρομή, ε, δημιουργία δυνατοτήτων και να εξετάζεται λίγο πιο προσεκτικά ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται οι συμφωνίες αυτές. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ και εσάς και το Πανεπιστήμιο του Κρόνιγκεν. Πολύ ενδιαφέροντα. Είμαστε εν αναμονή της ε, τελικής εκδοχής της μελέτης, το Μάιο αν άκουσα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφοι για τη συζήτηση. Πάμε στο σημείο 21 τώρα, διάφορα. Να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για την ε, στρατηγική της κυρίας ε, Μπεγκίν θα καθυστερήσει για αντί για 12 στις 21 Τετάρτου είναι 6 το απόγευμα στις 21 Τετάρτου. Τίποτα άλλο. Επόμενο σημείο, τελε... επόμενη συνεδρία 23 και 24 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ.